Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ να καθίσετε. Θα ξεκινήσει η συνεδρίαση. Και αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θα ξεκινήσουμε ευθύ αμέσως. Θα ήθελα μόνο να σημειώσω ότι στην Επιτροπή Άφετα αύριο έχουμε για το απόγευμα ένα σημείο σχετικό με τις συζητήσεις ε, ως προς την κοινοβουλευτική δουλειά στην ε, ασφάλεια και την άμυνα, σε σχέση με την κοινή πολιτική για την ασφάλεια και την άμυνα. Φροντίσαμε να περιληφθεί στην εμερική διάταξη για την αυρία συνεδρίαση, σε συνεργασία με την ΑΦΕΤ. Θα γίνει συζήτηση και για την εξωτερική υπηρεσία, εξωτερική δράση καλύτερα, αλλά και για το Κωσυφοπαίδιο και τη Βοσνία. Θα συζητηθούν οι εκθέσει. Έχουμε δύο αποστολέ και πάω. Δύο στη Βοσνία, μία στο Κοσμοπέδιο και γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα είναι ενδιαφέρουσε και για εσά. Και συνεδρία του Προεδρείου και των τονιστέ. Στο τέλο τη συνεδρίασή μα σήμερα. Σήμερα περιμένουμε, μάλλον έχουμε να υποδεχθούμε τον πρέσβευτή κύριο Κάρλο Φερνάντε Αρία, που προεδρεύει τη Ισπανική Προεδρία τη Εργασία του Συμβουλίου ως Ευχαριστούμε που ήρθατε κύριε Προσβευτά. Θα μας ε, παρουσιάσετε και θα συζητήσουμε δύο μεγάλες πτυχές. Θεσμική καταρχάς, με τη θέσπιση της Συνθήκης Λισαβόνας, τι αλλάζει και την ε, πτυχή που αφορά τις αποστολές της ε, ΚΕΠΑ. Σας δίνω το λόγο της αμέσως για να συνεχίσουμε με τη συζήτηση, παρακαλώ. Πρόεδρε, κύριε Τανζό, κάθε φορά που με προσκαλείτε εδώ στο Κοινοβούλιο, αισθάνομαι την ίδια μηχανία. Ποια γλώσσα να διαλέξω για να μιλήσω. Εάν ε, επιλέξω το πιο πρακτικό, θα πρέπει να επιλέξω τα αγγλικά. Εάν ε, επιλέξω το ορθότερο πολιτικό, ή πατριωτικό, μάλλον είναι το... θα έπρεπε να διαλέξω τα ισπανικά. Αλλά μια και θαυμάσω και τη γλώσσα του Μολιαρούς και είστε και εσείς Γάλλος, θα ξεκινήσω στα γαλλικά και ίσως μετά να συνεχίσω στα αγγλικά και ενδεχομένω να απαντήσω σε ερωτήσει των βουλευτών στα γαλλικά, τα αγγλικά, τα ισπανικά, ακόμα και στα γερμανικά αν το επιθυμείτε. Καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω τη μεγάλη χαρά που μου δίνει δυνατότητα να έρθω ενώπιον σας για να μιλήσω στην Επιτροπή, Υποεπιτροπή Αμήνας ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να σας μιλήσω για αυτά τα οποία αναφέρατε κι εσείς, δηλαδή καταρχάς τα θεσμικά ζητήματα που έχουν να κάνουν της ΚΕΠΑ, τα θερμικά ζητήματα λοιπόν της ΚΕΠΑ, αλλά και για να καταγράψουμε τις εξελίξεις ως προς τις διάφορες αποστολές και δράσεις. Δεν θα επεκταθώ σε όλες βέβαια τις αποστολές, αλλά σε αυτές που δεν θα αναφέρω ασφαλώς μπορώ να δώσω απαντήσεις αν υπάρχει ενδιαφέρον σε ερωτήσεις σας. Είπα και νωρίτερα ότι από την ΑΦΕΤ, όταν, ε, και το, είπα μάλλον όταν επισκέφθηκα και την ΑΦΕΤ, ότι έρχομαι εδώ ως εκπρόσωπος της ε, Επιτροπής Πολιτικής Ασφάλειας του Συμβουλίου. Αυτό λοιπόν όχι μόνο ως εκπρόσωπος της Ισπανικής Προεδρίας, αλλά και ως εκπρόσωπος και πρόεδρος της υποεπιτροπής αυτής εξ των ε, μελών της Επιτροπής αλλά και της Προέδρου της, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης κ. Σάστον. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν νομίζω που έχετε πρόεδρο στην υποεπιτροπή σας ε, από την, από την ομάδα μας υπ' αυτούς τους όρους. Νομίζω ότι μέχρι τώρα μόνο ως εκπρόσωποι της προεδρίας, της εκάστοτε προεδρίας έχουν έρθει οι προκατοχοί μου. Τώρα είμαι και ως προεδρεύων Ακόμη και αν δεν υπάρχει προεδρία του ΚΟΠΣ ουσιαστικά, δεν έχει ακόμη θεσπιστεί, υπάρχει βέβαια ο όρος αυτός, υπάρχει ο θεσμικό όργανο υπηρεσία εξωτερικής δράσης με στην συνθήκη, αλλά ακόμη δεν έχει τεθεί σε λειτουργία ο μηχανισμός, ώστε να διοριστεί ο εκπρόσωπός της. Και άρα, με βάση και τη συμφωνία που είχε η Ισπανική Προεδρία με την κυρία Άστον, την εκπροσωπώ εγώ σήμερα. Στο εξάμεινο λοιπόν αυτό της Ισπανικής Προεδρίας και στα θέματα της ΚΕΠΑ. Ε, δεν λέτε. Α, μάλιστα, στις ΚΕΠΑ λοιπόν. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλες προκλήσεις διαφόρων φύσεων, θεσμικές καταρχάς, πολιτικές αφετέρου, αλλά και θεσμικές προκλήσεις, γιατί ασφαλώς θα γνωρίζετε ότι όλες οι αλλαγές που έφερε η συνθήκη της Λισαβόνας και η θέση σε λειτουργία των διαφόρων οργάνων που προκύπτουν σιγά σιγά είχαν σαν αποτέλεσμα και για τη δική μας την υπηρεσία και τις εργασίες. Ε, σημαντικές αλλαγές και παρακολουθείτε εκ του σύνεκης και την παρουσία του υπατού εκπροσώπου και την, παρουσία, και την δυνατότητα μάλλον για άσκηση του δικαιώματος πρωτοβουλίας προκειμένου να ε, εκτελεστεί όπως πρέπει η εξωτερική πολιτική, ο ρόλος του σε σχέση με την υπηρεσία εξωτερικών σχέσεων και όλα αυτά βέβαια. Προφανώς υπήρξαν ε, και σημαντική ανατροπή ω προ την καθημερινή μας δουλειά. Αλλά σιγά σιγά ξαναβρίσκουμε το ρυθμό μας και κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε όλοι οι οργανισμοί, όργανα και θεσμοί να μπορούν να συνεχίσουν τη δουλειά τους απρόσκοπτα. Ξέρω ότι θα σας επισκεφθεί σε μερικές μέρες και ο Πολ Κρίστοφερσαν στην ε, ΑΦΕΤ, αύριο για να σας μιλήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες για τα διάφορα αυτά θέματα. Επίσης, Υπάρχει μια άλλη κατηγορία θεσμικών προκλήσεων από την ε, συνθήκη για τις οποίες δεν γνωρίζουμε αρκετά πράγματα όπου γίνεται λόγος για τη μόνιμη προσώπηση, όπου γίνεται λόγος από τη συνθήκη για τη ρήτρα αμοιβές ε, συνδρομής, όπου γίνεται λόγος για την αλληλεγγύη από τη συνθήκη, όπου όλα αυτά είναι θεσμοί, είναι ιδέες και έννοιες καινοφανείς, μένα που ενδεχομένως αποτελούν ε, νέα έκφανση μιας παλαιότερης έννοιας ή ιδέας, αλλά που πάντως χρειάζονται νέα ανάπτυξη, νέα εξέλιξη, τόσο προς τις ε, έννοιες αλλά και προς την πρακτική. Η Ισπανική Προεδρία εν προκειμένου προσπάθησε να οργανώσει σεμινάρια θεματικού χαρακτήρα που αναφέρονταν στις έννοιες, ε, τις ιδέες ε, και που αφορούσαν περισσότερο τεχνικούς ειδικού ε, πραγματογνώμονες μέσα από ένα brainstorming, μια ανταλλαγή απόψεων οδοτικές, ώστε να καταγραφούν οι παράμετροι εκείνες οι οποίες μπορούν να προσδιορίσουν αυτές τις ιδέες, τις έννοιες, για να υποβληθούν στην ύπατη εκπρόσωπο αυτές οι ιδέες για να ξεκινήσει την, τις ε, εργασίες της. Να μελετήσει δηλαδή, τις υποθέσεις αυτές και να προχωρήσει. Αυτά λοιπόν. Είναι πρόημα βέβαια να πούμε ότι ε, έχουν οριμάσει όλα αυτά. Πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση, η ανταλλαγή ιδεών και μεταξύ των κρατών μελών σε επίσημο επίπεδο και μεταξύ βέβαια και σε επίπεδο κοινοβουλίου ασφαλώς. θα μας απασχολήσουν λοιπόν και φέτος και στο πρώτο εξάμεινο του 2011 τουλάχιστον. Οι πολιτικές προκλήσεις επίσης είναι αυτές τις οποίες καθημερινά αντιμετωπίζουμε, αυτές που βλέπουμε καθημερινά στον τύπο και που προσδιορίζουν τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στις διάφορες περιοχές που δραστηριοποιείται, Επί παραδείγματι, στη Σομαλία, όπου έχουμε πολλά προβλήματα, όπω γνωρίζετε, έχουμε την Ατελάντη καταρχά στην αποστολή, έχουμε τα προβλήματα τη πειρατεία, αυτά που είδαμε ακόμη και χθε και σήμερα το πρωί στη Σομαλία, με ζητήματα τα οποία μας προξενούν ανησυχία φυσικά. Ξεκινήσαμε κάποιες δράσεις για να ενημερώσουμε την ε, μεταβατική ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Σομαλίας ώστε να προετοιμαστεί για να μηνθεί έναντι των δυνάμεων της Αρσαμπά, των Αταρτών. Ε, η UETN επίσης έχει ξεκινήσει μόλις τη δράση της αυτές τις ημέρες, θα σας μιλήσω διεξοδικότερα αργότερα. Μετά έχουμε τη Βοσνία που ε, εξακολουθεί να αποτελεί πηγή ανησυχίας. Προβλήματα πολιτικής αστάθειας. που εντείνονται και από τις επερχόμενες εκλογές. Στο τέλος του χρόνου έχουν προβλεφθεί. Έχουμε την Αλφαία, έχουμε την αστυνομική δράση, έχουμε την πολιτική μας ε, παρουσία εκεί με την προσπάθεια να διαφυλάξουμε την ομαλότητα, αλλά ξέρουμε ότι είναι όλο και πιο έντονη η διαλκυστίνδα μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων και τα πολιτικά κόμματα δεν καταφέρνουμε να τα επαναφέρουμε στην ομαλότητα όπως θα επιθυμούσαμε. Επίσης εμφανίζονται και νέες προκλήσεις αναπάντηχες, όπως ο σεισμός της ΑΕΤΗΣ, στον οποίο χρειάστηκε να δείξουμε ανταπόκριση, στην κρίση δηλαδή που προκάλεσε, όχι μόνο την ανθρωπιστική αλλά και την οικονομική κρίση, την ανοικοδόμηση δηλαδή με την προσφορά ε, μέσων, όχι μόνο των κλασικών εκείνων που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ανθρωπιστική βοήθεια, ταχεία ανταπόκριση, ανοικοδόμηση, αλλά και με στρατιωτικά μέσα προσφερθήκαμε. Τα κράτη-μέλη δηλαδή προσέφεραν τα στρατιωτικά τους μέσα με το συντονισμό μιας μικρής μονάδας επίπεδος ε, συμβουλίου, πράγμα το οποίο επέτρεψε στην, στα κράτη-μέλη, την Ένωση, να έχουν σαφέστερη και πιο ορατή παρουσία στην δύσκολη αυτή κατάσταση στην IT. Για πολλά θέματα, ασφαλώ η, Επίτροπο, η Υπουργός της Άμυνας, κυρία Τσακών, έχει έρθει στην Επιτροπή σα από την γνωρίζω, 4 Μαρτίου σας μίλησε. Αμέσως δηλαδή μετά την άτυπη σύνοδο στην ε, Μαγιόρκα, στην Παλμανή Μαγιόρκα των Υπουργών Άμυνας Πολλά από τα θέματα αυτά λοιπόν σας τα έχει παρουσιάσει η ίδια. Και από τότε, από 3 Μαρτίου, έχει συνέλθει μια φορά τακτικό συμβούλιο των Υπουργών των Εξωτερικών, με παρουσία και των Υπουργών Αμήνης, για ενημέρωση. Αν και θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν κοινό συμβούλιο, στις 26 Απριλίου στο Λουξεμβούργο. Και αν δεν απατώμε, ήρθε στην, Κούπερ, στην ΑΦΕΤ ο κύριος Κούπερ για να σας μιλήσει για ε, τα θέματα που απασχολούν τους υπουργούς των εξωτερικών στο Συμβούλιο. Να σας πω τώρα για την πλευρά των υπουργών αμήνης για τη σύνοδο αυτή. Πολύ σημαντικό και αυτό καταρχάς για την παραμονή μάλλον την Κυριακή 25 Απριλίου έλαβε χώρα, παρετέθη Δίνο μεταξύ της είπα της εκπροσώπου και των Υπουργών Αμήνης. Ήταν η πρώτη φορά δηλαδή που συναντούσε, είπατε, εκπρόσωπος ε, τους ε, υπουργούς, τους 27 υπουργούς αμήνης, γιατί μέχρι τώρα δεν είχε την ευκαιρία να ε, πάει. Δεν είχε πάει στην Πάρμαντα Μαγιόρκα, Φερρυπίν, τον Φεβρουάριο. Και άρα, ναι, ήταν άτυπημένη συζήτηση, πλην όμω πολύ ζωντανή, πολύ ενδιαφέρουσα. Έφυξε διάφορες θεσμικές πτυχές τη δυνατότητα να ενισχυθεί η ορατότητα στην ε, παρέμβαση των Υπουργών Αμήνης, να τους επιτραπεί ανεξαρτήτως και χωρίς ε, την παρουσία των Υπουργών των Οικονομικών να λαμβάνουν αποφάσεις για θέματα των αποκλειστικών τους αρμοδιοτήτων, όπως για θέματα δυναμικού, παραδείγματι, capacity ή άλλο. αντίστοιχα. Και ναι, αυτά τα μικρά συμβούλια, ε, κοινά δηλαδή συμβούλια άμυνας και εξωτερικών, είναι δύσκολο να ε, οργανωθούν, έχουν μια λεπτή χορογραφία. Μέχρι τώρα μάλλον ήταν κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Μπορούσαμε να έχουμε παράλληλη προεδρία από έναν Υπουργό Αμήνης και έναν Υπουργό Εξωτερικών, δύο παράλληλων συμβουλίων που ολοκλήρωναν τη δουλειά τους για να συνέλθουν μετά από κοινού. Ωστόσο τώρα βλέπουμε ότι γίνεται μια διαδοχική μάλλον συνεδρίαση και μετά υπάγονται όλα αυτά στο Συμβούλιο, αυτά τα θέματα που θα έχουν καλύψει Υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών, στο ε, ε, Υπουργείο στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Πάρα πολλή δουλειά και κυρίως για την κυρία Άστον. Ήταν μια πολύ σκληρή μέρα αυτή στο Λουξεμβούργο για την ίδια. Και πρέπει βέβαια να ε, επιδειχθεί και ιδιαίτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα στο να διακριθούν τα ζητήματα που θα απασχολήσουν τα συμβούλια, στο να επιλεγούν τα θέματα στα οποία είναι απαραίτητο να είναι παρόντε και οι Υπουργοί Εξωτερικών και οι Υπουργοί Αμήνη, μετά για κάποια άλλα θέματα που θα πρέπει να συνεδριάζουν και να συζητούν χωριστά. Όλα αυτά συζητήσαμε. Συζητήσαμε επίσης πώς οι πολιτικο-στρατιωτικές πτυχές, δηλαδή πτυχές διαχείρισης κρίσεων, θα ενσωματώνονται, θα ενσωματωθούν μάλλον στις δομές της εξωτερικής υπηρεσίας. Έδωσε η κυρία Άστον κάποιες γενικές ιδέες, εξηγώντα ταυτόχρονα και τις εξελίξεις στην υπόθεση αυτή. Συζητήθηκε επίσης το πώς μπορούμε να, ή τι είδους διδάγματα μπορούμε να αποκομίσουμε από την ε, κρίση της IT, πώς πρέπει να βελτιωθεί η ανταπόκριση ταχεία και ε, πλήρης ανταπόκριση σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και άλλων κρίσεων. Τα battle groups επίσης, οι ομάδες κρούσεως, ή εκτός αυτών οι ομάδες συντονισμού όπως αυτή της ITs πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή αν χρειάζεται μια μόνιμη μονάδα ή μια μόνιμη δομή καλύτερα για να μας βοηθάνε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Άρα το δείπνο είχε πάρα πολύ ψητό. Πολύ ουσία. Και ήταν και η πρώτη φορά που συνάντησαν την επατρική πρόσωπο Υπουργεία. Η υπόλοιπη συνεδρίαση ακολούθησε τη συνήθη δομή. Οι Υπουργοί τη Αμήνας συζήτησαν για το δυναμικό, για την ε, ασφάλεια των θαλασσιών μεταφορών, ιδιαίτερο ανταπόκριση στην κρίση. Τι συζητήσαμε τις διάφορες ε, δράσεις και μετά έγινε και μία κοινή συνεδρίαση μαζί με τους Υπουργούς Εξωτερικών για το Αφγανιστάν και παρουσία του κ. Ράσμουσεν, προσώπου του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ. Αν και νομίζω ότι ο κύριος Κούπερς τα ε, εξέθεσε όλα αυτά. Γιατί εκεί έκλεισαν συνεδριάσεις με ε, έγκριση από τους υπουργούς ε, των θέσεων αυτών για την ε, εξωτερική για την ασφάλεια και την ε, ε, θαλάσσια ασφάλεια. Ευχαριστώ και τώρα στα αγγλικά. Θα ήθελα να σας εξηγήσω. Να σας δώσω κάποιες ιδέες σε σχέση με τις ε, πολιτικο-στρατιωτικές ε, επιχειρήσεις. Θα ήθελα να σας ε, αναφέρω καταρχήν και αναφέρω και προηγουμένως την Βοσνία. για την επιχείρηση Αλτία. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ότι αυτή η επιχείρηση ήταν επιτυχή όλα αυτά τα χρόνια, γιατί διατήρησε ένα σταθερό περιβάλλον στην Βοσνία όσον αφορά τον τομέα της ασφάλειας και πιστεύω ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει επιτυχή σε αυτή η επιχείρηση όσο ακόμα χρειάζεται να λειτουργήσει. Έχουμε τώρα την πρόκληση των εκλογών στα τέλη του χρόνου και αποφασίσαμε να διατηρήσουμε την επιχείρηση αυτή σε ένα μίνιμουμ ε, επίπεδο ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί μέχρι τουλάχιστον μετά τις εκλογές και θα δούμε αργότερα ποιο μέλλον θα έχει. Ταυτόχρονα αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τη νέα επιχείρηση Αλθεία που είναι μία μη εκτελεστική αποστολή, δηλαδή ε, θα παρακολουθεί και θα συμβουλεύει καθώς και θα καταρτίζει το στρατό της Βοσνίας. Κάτι το οποίο ήδη γίνεται, αλλά πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό έργο και πρέπει να συνεχιστεί. Όσον αφορά το εκτελεστικό τμήμα, το βασικό πρόβλημα ήταν αν μπορούσαμε να διατηρήσουμε όλα αυτά τα εκτελεστικά κομμάτια μέσα στο πλαίσιο της αποστολής, γνωρίζοντας ότι πολλά κράτη-μέλη έχουν επαναφέρει τον κόσμο. Και η αποστολή σιγά σιγά άρχισε να έχει ελλείψεις. Ο στρατηγός Μπολτ που είναι επικεφαλής της αποστολής, έχει εξασφαλίσει το απαραίτητο επίπεδο στρατευμάτων μέχρι το τέλος του έτους. Γιατί υπήρξαν ταυτόχρονα κάποια κρατημέλη τα οποία αύξησαν την συμμετοχή τους για να καλύψουν τα κενά και να μπορέσει να διατηρηθεί το ίδιο επίπεδο στρατευμάτων. Είμαστε ευγνώμονες στην Αυστρία που που έστειλε έναν επιπλέον λόγο και ελπίζουμε να αποφύγουμε περαιτέρω περικοπές ε, φέτος γιατί διακυβεύεται η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, μετά το 2010 και υπό το φως των τελευταίων συμπερασμάτων του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων είδαμε, ε, αποφασίστηκε ότι θα επανεξεταστούν αυτές οι επιχειρήσεις, να θα διατηρηθεί η βοήθεια για την ε, αεροπορία Ε, και τα κράτη-μέλη φαίνεται να έχουν τη δυνατότητα και την βούληση να διατηρήσουν ε, στα ίδια επίπεδα ε, τις στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται επί τόπου. Αυτό θα συζητηθεί βέβαια σε αυτό το χρόνο αφού θα ληφθεί υπόψη και το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο. Τώρα, σε σχέση με με την Αταλάντη, που είναι μια σημαντική και επιτυχής επίσης επιχείρηση, αποστολή. Το είχαμε, έχουμε να, να εξαλείψουμε το πρόβλημα των, της πειρατείας στον Ειδικό ωκεανό. Έχουμε καταφέρει έναν μεγαλύτερο βαθμό ασφαλούς περιβάλλοντος στον κόλπο του Άντεν και στη ανοιχτά της Σομαλίας. Η επιχείρηση Αταλάντη κατάφερε να προσφέρει προστασία στα ειδικά σκάφη που δίνουν βοήθεια στη Σομαλία ε, ώστε να δώσουν επίσης ε, τα φορτία τους ε, στην ε, ειρηνευτική αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία, καθώς και να δώσουν βοήθεια και προστασία στα ευάλωτα σκάφη, όπως τα αποκαλούμε, δηλαδή εμπορικά σκάφη, αλλιευτικά σκάφη, σκάφη αναψυχής και ούτω καθεξής. Το να διακοπούν οι πειρατικές αυτές ε, δραστηριότητε ε, θέλουμε να το καταφέρουμε όχι μόνο στον ε, διάδρομο του κόλπου του Άντεν αλλά και στις, στη λεκάνη της Σομαλίας. Υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία συμμετέχουν στην επιχείρηση Αταλάντη, Νορβηγία και η Κροατία και δύο νέα που θέλουν να συμμετέχουν σε λίγο καιρό δηλαδή Ουκρανία και ε, Μαυροβούνιο. Και αυτό αποδεικνύει το ενδιαφέρον και την επιτυχία της επιχείρησης. Αυτό όχι μόνο μέσα στο πλαίσιο της επιχείρησης Αταλάντη, αλλά και σε συνεργασία με αυτή την επιχείρηση έχει εκφραστεί μεγάλο ενδιαφέρον από τρίτα μέρη. Υπάρχει πολύ καλό συντονισμός και συνεργασία με το ΝΑΤΟ. ιδιαίτερα αποτελεσματικό λόγο του SHADE, δηλαδή κοινή ενημέρωση και επίλυση ε, κρίσεων, συνοντονισμός δηλαδή μεταξύ όλων των δυνάμεων που ενεργούν ε, στην περιοχή. Οι Κινέζοι ε, εντωμεταξύ είναι όλο ένα και πιο δραστήριοι και έπρεπε να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Αποστολή, ιδιαίτερα αναλαμβάνοντας ευθύνη σε κυλιόμενη βάση εκπεριτροπής για να βοηθήσουν στον έλεγχο του διεθνούς ε, διαδρόμου στον κόλπο του Άντεν. Το ρωσικό ναυτικό επίσης ε, είναι σε συντονισμό με την επιχείρηση Αταλάντα, Αταλάντη. Το δεύτερο τμήμα που είναι κάπως πιο ανησυχητικό είναι αυτό που αφορά την κράτηση και τη δίωξη των ε, υπόπτων πειρατών και θα γνωρίζετε πολύ καλά ότι μέχρι, σε αυτή, τη, μέχρι αυτή τη στιγμή η Κένια έκανε τη μεγαλύτερη συνεισφορά και οι Σεϊχέλες επίσης. λήφθη απόφαση από τις αρχές της Κένιας ότι θα ήθελαν να, να σταματήσουν τις συμφωνίες μεταφοράς. Υπήρξαν κάποιες, δημο, κάποια διπλωματικά διαβήματα που έγιναν στις 23 Απριλίου. Ατύπως ε, καταγράφηκε ότι ο πρόεδρος θέλησε να αντιστρέψει την απόφαση και ότι έγινε μια υπουργική μάλλον έχει προγραμματιστεί μια νέα υπουργική διάσκεψη για να εξεταστεί αυτό το θέμα, δηλαδή σε λίγες μέρες. Ο ύπατος εκπρόσωπος ε, αποφάσισε να στείλει τεχνικές ε, αποστολές, η μία αφεύγει αύριο νομίζω και θα βρίσκεται επί τόπου κάπου τον Μάιο, όχι για να συνομιλήσει μόνο με την κυβέρνηση της Κένιας, αλλά και με τις άλλες πέντε χώρες με τις οποίες συνομιλούμε, ώστε να, έχουμε, να συνάψουμε κάποιες ε, συμφωνίες ε, με τα, με, μεταφοράς ε, Μαυρίκιος, Μοζαμβίκη, Τανζανία, Ουγκάντα, εκτός από τις Αιχέλες που σας ανέφερα προηγουμένως. Αλλά δεν θα σταματήσει ο κατάλογος εδώ. Θα σκεφτούμε και άλλες δυνατότητες σε άλλες χώρες και θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε την φαντασία μας. Αυτά για την επιχείρηση Αταλάντη. Φυσικά η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να στηριχτεί αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα στην περιοχή και γι' αυτό ανέφερα το UTM Σομαλία, η οποία έχει φτάσει στην αρχική της ε, ε, επιχειρησιακή ικανότητα στις 23 Απριλίου και ο επικεφαλής της αποστολής είναι έτοιμος να αρχίσει να εργάζεται από την 1η Μαΐου. Τα πάντα εξαρτώνται από την μεταφορά των πρώτων ε, εκπαιδευομένων στο στρατόπεδο Χουγκάντα. Τα στρατηγία στην Καμπάλα έχουν ε, φτιαχτεί, καθώς επίσης υπάρχει και μια ανταπόκριση στο Ναϊρόμπι και εδώ στις Βρυξέλλες μια άλλη. Ε, είναι έτοιμη δηλαδή η αποστολή, είναι έτοιμη να αρχίσουν την κατάρτιση, την εκπαίδευση μόλις θα έχουν φτάσει οι, εκπαιδευόμενοι. Εμείς ε, θέλουμε να προσφέρουμε ε, ειδικά μόντουλ για όλους τους εκπαιδευόμενους. Όταν λέμε μόντουλ θα πει διάφορα ειδικά ε, ειδικού εξοπλισμού για το τι μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν οι στρατιώτε εκεί. Δηλαδή, πόλεμο σε αστικές περιοχές, ε, η ειδική εκπαίδευση σε σήματα, σε ιατρικές ειδικεύσει, δημιουργία πνεύματο ομάδας σε μικρές μονάδες που μπορούν να ε, πολεμήσουν σε επίπεδο μικρών ομάδων. Και η ιδέα είναι να αναπτυχθεί επίσης κάτι το οποίο ίσως να μην χρησιμοποιείται σε εκείνο το μέρος του κόσμου, δηλαδή η ιδέα μιας μονάδας ε, πολύ ενωμένης μεταξύ της και η εξάμενη εκπαίδευση θα αφιερωθεί σε αυτό. Θα ολοκληρωθεί η αποστολή το 2011 το Μάιο, αφού θα έχουν γίνει δύο εξάμενα εκπαίδευσης και θα έχουν εκπαιδευτεί 2.000 στρατιώτες για λογαριασμό της ομαλικής κυβέρνησης. Αυτές είναι οι τρεις κύριες αποστολές. Να πω κάτι για μια πολιτική αποστολή. Δεν θα μιλήσω πολύ περισσότερο γιατί προτιμώ να ακούσω δικές σας ερωτήσεις, αλλά να σας πω δύο λόγια για το Αφγανιστάν που ξέρω πως σας ενδιαφέρει πολύ. Συζητήθηκε το Αφγανιστάν τον Απρίλιο μεταξύ των Υπουργών Αμήνης και Εξωτερικών Υποθέσεων και του ΝΑΤΟ. Η U-Poll είναι ένα βασικό κλειδί για την, ε, όσον αφορά την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της κρίσης στο Αφγανιστάν. Η αποστολή ξεκίνησε το 2007, ξεκίνησε με πολλές δυσκολίες, αλλά τώρα προοδεύει στην εφαρμογή της εντολής της. 300 άτομα είναι το προσωπικό Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να μας απασχολούν τόσο οι αριθμοί, τα αριθμητικά στοιχεία, αλλά το τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, η Ιούπολ θέλει να κάνει μια συγκεκριμένη συμβολή όσον αφορά την ε, πολιτοφυλακή, που είναι μια ένα συμπλήρωμα για, την, για το Αφγανιστάν. Είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που κάνει το ΝΑΤΟ με τη δική του εκπαιδευτική αποστολή στο Αφγανιστάν. Εκπαιδεύει ε, το ΝΑΤΟ απλούς ανθρώπους για να γίνουν στρατιώτες. Η UPOL κάνει συγκεκριμένη εξάσκηση στους αστυνομικούς ώστε να μάθουν διάφορες τεχνικές όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, τις έρευνες, ε, την κατασκοπία, ε, την καθοδήγηση οργανωτικούς και δηλαδή είναι ένα συμπληρωματικό έργο που συνδέεται πολύ περισσότερο με τις ανάγκες του, δημιουργία της δημιουργίας κράτους δικαίου από πλευράς της αφγανικής κυβέρνησης και όχι, δεν έχει στόχο το να δημιουργηθούν αστυνομικές δυνάμεις στο Αφγανιστάν. Συνεχίζεται η εργασία εκεί. Ε, ίσως να γίνει μια επέκταση και προσαρμογή τη εντολή. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να εξετάσουμε την ανάπτυξη της UPOL στις διάφορες επαρχίες, ίσως και να εγκαταλείψουμε κάποιες από αυτέ, αλλά να ενισχύσουμε άλλε ταυτόχρονα. Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς θα συνεργαστούμε καλύτερα με τον ΝΑΤΟ και αυτό συζητήθηκε ευρύτατα στο Αφγανιστάν. Τώρα δεν ξέρω πώς είμαστε από χρόνο, αλλά δεν θέλω να μακρηγορήσω για να υπάρξει χρόνος και για ερωτήσεις και για συζήτηση. Ίσως λοιπόν να σταματήσω τώρα. Αν κάτι δεν ανέφερα, δεν σημαίνει πως ε, δεν θα απαντήσω, εάν με ρωτήσετε γι' αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη. Ακριβώς αυτό είναι και η σκοπιμότητα δούμε να μπορέσουμε να ακούσουμε τα θέματα που σας απασχολούν ε, στην, ε, εξωτερική, στην υπηρεσία εξωτερικών σχέσεων. Θα παρακαλέσω και τους συναδέλφους να λάβουν το λόγο. Και θα ήθελα και εγώ βέβαια να ακούσω τι έχει να μας πείτε για τέτοια θέματα. Την πρώτη αυτή συνεδρία με την κυρία Αστόν, καταρχά στο Λουξεμβούργου. Τι γίνεται σε σχέση με την ε, λεγόμενη μόνιμη αντιπροσωπεία που δεν έχει πολύ σωστή εικόνα, ορισμούς, ε, περιμέτρους, ουσία και επίσης να το Ευρωπαϊκή Ένωση. Μίλησατε για την παρουσία του Ράσμουσεν στην ε, συνεδρία σε αυτή. Επίσης η κυρία Άστον έχει πολλές φορές επισημάνει ότι έχει αγαθές σχέσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Πλην όμως παραμένουν ε, σε ορισμένα θέματα, προβληματικές αυτές οι σχέσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συνεργασία στο Αφγανιστάν, για το Κόγκο που ίσως δεν είναι πια τόσο ε, επικίνδυνο, μπορούμε να περιμένουμε μια ε, πιο απρόσκοπτη συνεργασία, αλλά το Αφγανιστάν σίγουρα έχει άλλους, άλλες παραμέτρους. Επίσης αναφερθήκατε στην Αλθέα, την επιχείρηση Αλθέα. Ποια είναι η αξιολόγηση της πραγματικής κατάστασης εκείνη η οποία υπαγορεύει τη διατήρηση στρατιωτικής παρουσίας. Ναι, η πολιτική κατάσταση μπορεί να είναι δύσκολη στη Βοσνία, αλλά είναι διαρθρωτικά δύσκολη ε, και θα παραμείνει δύσκολη για πολλά χρόνια από ό,τι βλέπουμε και για λόγους εκλογικών αντιπαραθέσεων και για λόγους ε, ε, πολιτικού λόγου εθνικιστικού που επιλέγουν κάποιοι. Εν πάση περιπτώσει δεν βλέπω στρατιωτικά ποιο είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να διατηρηθούν ποια είναι η ανάγκη για την προστασία της ασφάλειας, της φύλαξης ασφάλειας και της τάξης πέραν της συμβολικής βέβαια παρακολούθηση πολιτικής διαδικασίας συμφιλίωσης ε, στην περιοχή αυτή. Ε, αυτές οι δικέ μου Ο κύριος Πασκού παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέσβη για την ενημέρωσή σας. Δύο ερωτήσει έχω. Η μία είναι γενικότερη, η άλλη είναι κάπως πιο εξειδικευμένη. Η πρώτη, θα ήθελα να μου πείτε αν υπήρχε κάποια πρόθεση, αν υπάρχει πρόθεση να εμπλακούν στη διαδικασία των συμπερασμάτων μαθημάτων μετά από την έκρηξη του ηφαιστείου στην Ισλανδία αυτή η διάσταση της άμυνας και της ασφάλειας με κάποια ειδικά μέτρα για αντιμετώπιση κατεπήγοντος ή κάτι παρόμοιο. Αν είναι κάτι, αν υπάρχει κάτι το οποίο ακολουθείται παράλληλα με αυτή τη γραμμή. Το δεύτερο αφορά την Βοσνία Ζεγοβίνη αυτό. Θα έλεγα ότι εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε μεταξύ την διοργάνωση και την λειτουργία σε σχέση με Υπουργεία Άμυνα και στρατιωτικέ δομέ, πράγμα το οποίο είναι παλαιό πρόβλημα βέβαια. Αλλά είπατε ότι επίση υπάρχουν υποστηρικτικέ δράσει που παρέχονται. Θα ήθελα να μου πείτε πού τίθεται το κέντρο βάρου σε αυτέ τι δράσει. Είναι θεσμικέ δράσει ή είναι στην κατάρτιση και εκπαίδευση προσωπικού. Για να μην ξεχνάμε ότι είναι μια γενεά η οποία τώρα εξαλείφεται σε σχέση με την ε, πραγματική εμπειρία, η πείρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρος κ. Λίζεκ. Για να δυσκολέψω τα πράγματα θα κάνω την ερώτησή μου στα πολωνικά. Panie Ambasadorze, ε, ε, jestem... Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρέσβη, έχω την εντύπωση ότι προσπαθήσατε με συμπυκνωμένο τρόπο να δώσετε μία σύνοψη, μία περίληψη όλων των δραστηριοτήτων σε αυτούς τους τομείς όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, όλων όσων εξελίσσονται σε αυτό το επίπεδο. Αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρον θα έλεγα είναι σίγουρα η δομική, η διαρθρωτική πτυχή σε σχέση με αυτά τα οποία αναφέρατε. Λοιπόν, σε σχέση με αυτό, κάτι πολύ συγκεκριμένο που αφορά την Ευρωπαϊκή Διπλωματική Υπηρεσία, την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Έχει μεγάλη σημασία νομίζω. Θα ήθελα το εξή ερώτημα να διατυπώσω. Θα ήθελα να μου πείτε τι γίνεται σε σχέση με το όραμα της Προεδρίας. Γνωρίζω φυσικά ότι είναι μια ανακυκλούμενη, ένα αλλάξει Προεδρία. Έχουμε τώρα δύο μήνες ακόμα που θα διαρκέσει η Ισπανική Προεδρία. Θα ήθελα να μου πείτε τι γίνεται με τις σχέσεις με τους Υπουργούς Εξωτερικών και τους Υπουργούς Άμυνας μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Με άλλα λόγια, γνωρίζω τι γίνεται όταν οι Υπουργοί Άμυνας συναντώνται χωρίς τους Υπουργούς ε, Εξωτερικών και τα λοιπά, εντάξει για κάποιες φιλοδοξίες ε, που εκφράζονται και θέλουν να καλύψουν. Αυτό επιθυμούν οι Υπουργοί Άμυνας, δηλαδή επιθυμούν το δικό τους ε, θεσμικό όργανο να έχει περισσότερες αρμοδιότητες θα έλεγα στον τομέα της άμυνας. Όταν όμως συνεδριάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών χωρίς τους Υπουργούς Άμυνας, κάπως διαφορετικά έχουν τα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, το αντίθετο δηλαδή συμβαίνει σε σχέση με τη συνάντηση των Υπουργών ε, Άμυνας. Όταν συναντώνται από κοινού, ε, τότε τι συμβαίνει. Μάλλον στο δείπνο επικεντρώνονται στο οποίο αναφέρατε. Πώς αντιμετωπίζει η Ισπανική Προεδρία αυτό το πρόβλημα. Πώς σκέπτεται να επιλύσει αυτό το πρόβλημα σε αυτές τις σχέσεις ή αυτές τις τριβές που υπάρχουν. Και μια πολύ εξειδικευμένη ερώτηση ε, όσον αφορά τη γεωργία είναι σε όλους μας σαφές ότι στην Γενέβη διεξάγονται συζητήσεις και διαβουλεύσεις για το ζήτημα της γεωργίας. Δεν θέλω όμως να μου πείτε αν εσείς μπορείτε να φανταστείτε ότι στο μέλλον για παράδειγμα, μελλοντικά, κάποιες διεθνείς ε, αμυντικές δυνάμεις, ένοπλες δυνάμεις, ιδιαίτερα ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην Απχαζία για παράδειγμα και στη Βόρεια Οσετία Μπορεί αυτό να γίνει, δηλαδή η πιθανότητα, ε, α ας το πω έτσι, συνεργασίας των Ευρωπαϊκών Ενόπλων Δυνάμεων και συνεργασίας με τις ρωσικές δυνάμεις. Τι είναι δυνατό να γίνει και πώς μπορεί αυτή η δυνατότητα να εξελιχθεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Πρέσβη για αυτή την ευρεία. Δηλαδή, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μας ε, παρουσιάσατε διάφορες πτυχές ε, της ε, κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής μάλλον ασφάλειας και άμυνας. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Ε, καταρχήν ε, θα ήθελα να βάλω μια ερώτηση στον πρόεδρο Τανζάν σε σχέση με την συζήτηση για την ε, δομημένη συζήτηση. Και μάλιστα η πρώτη μου ερώτηση αφορά μία δομένη συνεργασία ή τις δομένες συνεργασίες και γενικότερα πώς σκοπεύετε να συνδυάσετε από τη μια πλευρά την απαραίτητη φιλοδοξία του αντικειμένου δηλαδή της δεδομένης συνεργασίας ε, από μόνιμη, ιδιαίτερα από, υπό το προφίλ της ανάπτυξης δυνατοτήτων και των επιχειρησιακών ε, δυνατοτήτων και από την άλλη πλευρά το στοιχείο της, ε, του, ανοιχτού, του, του ανοιχτού της χαρακτήρα και η δεύτερη ερώτηση, κάνατε μια ερώτηση πολύ ενδιαφέρουσα σε σχέση με το αν θα μπορούσε να καταστεί σταθερό, σταθερή η μονάδα συντονισμού που συντόνισε την αποστολή στρατιωτικών μέσων στο πλαίσιο του ΟΗΕ στην IT. Ε, Διερωτώ αν υπήρξε και πώς λειτουργήσε ο συντονισμός ανάμεσα σε αυτή τη μονάδα συντονισμού και τις εργασίες συντονισμού σε πολιτικό επίπεδο, όπως αυτές έγιναν από την MIC στο πλαίσιο του κοινοτικού μηχανισμού για την ε, πολιτική προστασία και αν πιστεύετε ότι στο μέλλον αυτές οι δύο πτυχές συντονισμού της χρήσης δηλαδή στρατιωτικών μέσων για την πολιτική προστασία και το συντονισμό των δραστηριοτήτων που είναι καθαρά πολιτικού χαρακτήρα, πώς μπορεί να συνεχιστεί και πώς μπορούν αυτά να συνδυαστούν σε σχέση με τον ρόλο που θα παίξει και η εξωτερική υπηρεσία σε αυτό το πλαίσιο. Και επίσης, η το κείμενο του Συμβουλίου κάνει μια αναφορά στη διεύθυνση διαχείρισης κρίσης και σχεδιασμού, που είναι σίγουρα μια θεμελιώδης δομή που θα πρέπει να εφαρμοστεί και να ε, οικοδομηθεί και στο πλαίσιο του σχεδίου δομής που θα έχει αυτή η υπηρεσία, πώς θα λειτουργήσει ο συντονισμός ανάμεσα σε αυτή τη δομή και τις άλλες ε, δομές, δηλαδή όπως η CPCC, αφού από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρχει μία διεύθυνση απάνω από αυτές τις ε, διάφορες υπηρεσίες. Θα είναι ο... Δεν θα αναφέρονται στο Γενικό Γραμματέα που ε, γίνεται πλέον εκτελεστικό όργανο, αλλά στην ΕΠΑΤΗ εκπρόσωπο. Τέλος, να σας πω ότι είναι ανησυχητικά εκεί η εξέλιξη Σομαλία, όχι μόνο η απόπειρα στην, στο αλλά και ε, η κατάληψη μιας βάσης επιρατών. αν υπάρξει σύγκρουση ανάμεσα στην ε, Σαμπάμπ Ισλάμ και ε, αυτή η κατάληψη φαίνεται να, να έχει γίνει ε, ως μια αντίδραση στην πειρατεία για λόγους προπαγάνδας ε, ή μήπως προκύπτει από την ανάγκη απόκτησης μιας πλουτοπαραγωγικής πηγής όσον αφορά την αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο αυτές περιοχές. Πώς εντάσσονται όλα αυτά στην αντιμετώπιση της Σομαλίας και πώς συνδυάζονται και με αυτή τη νέα στρατιωτική αποστολή, μάλλον ε, αποστολή εκπαίδευση στρατιωτικών στην Ουγγάντα. Ευχαριστώ πολύ. Thank ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρέσβη, μας δώσατε αρκετά ευρύ πλαίσιο για το πού πολεμάμε και διεξάγουμε τους πολέμους μας και προσπαθούμε να είμαστε παρόντες και να παρέμβουμε παγκόσμια. Αν θα το διατύπωνα λιγότερο διπλωματικά, θα έλεγα, μια και ήμουν επί πολλά χρόνια διπλωμάτης και τώρα έχω διαφορετικό καθεστώς, θα έλεγα ότι έχουμε υπερβολικό εύρος ανάπτυξης δυνάμεων και δραστηριοτήτων στον κόσμο. Φτάνουμε στα όρια μας φτάνουμε στα, στον ορισμό του παγκόσμιου χωροφύλακα σχεδόν θα έλεγα με όλα αυτά. Και αυτό θα μπορούσε να αληθεύει ή να είναι ακόμα πιο αληθές αν και αν, δεν υπάρχει μια σαφέστατη πολιτική ανάλυση και πολιτική στοχοθέτηση για το τι προσπαθούμε να κάνουμε και για το πώς θα θέλαμε να πετύχουμε αυτές τις δράσεις και να μπορέσουν αυτές οι δράσεις μας να στεφθούν με επιτυχία. Αυτό που είδα λοιπόν να λείπει στη δική σας αξιολόγηση είναι αυτό το στοιχείο. Μια πολιτική ανάλυση δηλαδή αυτών των δράσεων. Όλων αυτών των αποστολών δηλαδή. Των, της πληθώρας αποστολών που α, αναπτύσσουμε. Παράδειγμα, Βοσνία και εδώ σε σχέση με τα θέματα, οι ζητήματα που ε, ο πρόεδρος παρουσίασε και παρενέβη για τη Βοσνία ε, Ζεγοβίνη. Αληθεύει. Δεν είναι μόνο σημαντικό να έχουμε αρκετέ δυνάμει, αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζουμε γιατί υπάρχουν αυτέ οι ένοπλε δυνάμει εκεί. Δικαιολογείται η παρουσία του ε, σε σχέση με του στόχου. Είχα πάει στη Βοσνία Ζεγοβίνη αρκετέ φορέ. Μίλησα, είχα έτσι επαφή με πολιτικού και άλλου. Δεν θεωρούν ότι υπάρχει απειλή σε σχέση με την ασφάλεια στη Βοσνία Ζεγοβίνη, ώστε να δικαιολογείται έτσι μια σε τέτοιο εύρος ε, στρατιωτική παρουσία και αστυνομική παρουσία από την Αλοδαπή. Έχουν πολιτικά λοιπόν προβλήματα, εντάξει, και πολύ λιγότερο ε, επιτυχία, λιγότερη επιτυχία σημειώνουμε ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τους όσον αφορά το πολιτικό επίπεδο. Το πολιτικό και τα πολιτικά θέματα στη Βοσνία ξεκινούν απλά με το γεγονός ότι τα παιδιά, για παράδειγμα, πάνε σε ένα σχολείο και χρησιμοποιούν τρεις διαφορετικές εισόδους. Δεν μιλάνε το ένα παιδί με το άλλο όταν είναι από διαφορετικές κοινότητες. Έχουν διαφορετικά σχολικά βιβλία για την ίδια την ιστορία της πατρίδας τους. Και η νέα γενναία αναζωπυρώνει το μίσος και σε σχέση με, την, ε, με, τα παλαιά αίτια των, ε, του μίσους από την προηγούμενη γενναία. Θα πρέπει εδώ να δούμε αυτό το θέμα σε σχέση με την παρουσία μας εκεί με τις δυνάμεις μας ε, προσπαθώντας να ενισχύσουμε την κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια αλλά μόνο δικαιολογείται κάτι τέτοιο αν αλλάξουμε αυτά τα πράγματα και κατανοήσουμε τους όρους της πολιτικής αντιπαράθεσης και των πολιτικών προβλημάτων εκεί. Το ίδιο θα έλεγα ισχύει και σε μια διαφορετική δομή αλλά με και διαφορετικό τρόπο αλλά είναι το ίδιο πάλι πρόβλημα και στη Σομαλία. Μοιάζει καμιά φορά <clears throat> σαν μια ιδέα να έχει αναπτυχθεί σε ένα παιχνιδάκι, σε ένα κρυφτούλι μεταξύ πολεμικών πλοίων από δικών μας πλοίων φρεγατών και κορβετών και πειρατικών πλοίων, ποιος θα είναι πιο ε, αποτελεσματικός στη δράση, μακροπρόθεσμα τι γίνεται. Βλέπουμε να υπάρχει κάποιο φως στην άκρη της σύραγγας, στο τέλος της σύραγγας. Ξέρουμε τι προσπαθούμε να πετύχουμε και τι θα γίνει στο τέλος, τι θα επιτευχθεί ή όχι αντί να έχουμε μια τέρμονα αλλαγή και ιστοδιειναικές αλυσίδα αποστολής νέων ενόπλων δυνάμεων, προσκαλώντας νέες χώρες και ένοπλες δυνάμεις από αυτές να συμμετάσχουν και να αποσταλούν εκεί. Και τι συμβαίνει. Απλά ικανοποιούμαστε όταν κάποιοι, κάποιες νέες χώρες ε, λένε ότι είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν και να αποστείλουν δυνάμεις. Εκεί θα έπρεπε περισσότερο να μπορέσουμε να κάνουμε, περισσότερα να πετύχουμε με λιγότερη θα έλεγα παρουσία σε ενόπλες δυνάμεις εκεί. Γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι βέβαια μια πολύ ακριβή σαφής ερώτηση. Ζητώ συγγνώμη για αυτό τον άναρχο τρόπο διατύπωσης αυτής της ερώτησης ή του προβλήματος που θέτω με το ερώτημά μου αυτό. Αλλά είναι ουσιαστικό αυτό για την πολιτική που θέλουμε εμείς ως μέλη του Ευρωκοινοβουλίου να πετύχουμε. Ευχαριστώ. Merci, Σας ευχαριστώ κύριος Γκάλερ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Γκαρτιέρη, δύο από τα θέματα που ήθελα να θίξω τα ανέφερε ο ίδιος. Την CMPD και την Ουγγάντα επίσης. Και εγώ θα μπορούσα με γλαφυρό τρόπο να αναφερθώ σε κάποια θέματα όπως ο συνάδελφος Βάγγελ, όμως πιο εξειδικευμένα να αναφερθώ στο θέμα της CMPD και να ε, το θέσω πιο ε, εξειδικευμένα. Τα δύο εναλλακτικά οργανογράμματα, αν τα δει κανεί ε, σε σχέση με το Συμβούλιο για την Εξωτερική Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και όταν δει κανεί ε, και την ε, δεύτερη εναλλακτική λύση, CNPD και τις δύο άλλες μονάδες και σε σχέση με την είπα το εκπρόσωπο ε, του Συμβουλίου και είπα το εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική και έχουμε και την εναλλακτική δυνατότητα του Κοινοβουλίου ας το πω έτσι και της Γενικής Γραμματείας σε σχέση με την εξωτερική δράση και τη δομή. Θα μπορούσατε να μας πείτε γιατί το Συμβούλιο έχει αυτή την άμεση δέσμευση, ας το πω την οποία προτιμά και προωθεί και δεν επιλέγει την ε, διασύνδεση υπό τον έλεγχο ε, της Γενικής Γραμματείας. Όσο αφορά την Αταλάντη, πολλά θετικά πράγματα αναφέρθηκαν. Ξέρουμε όμως ότι η λύση για το ε, πρόγραμμα Αταλάντη βρίσκεται στην ξηρά, στη στεριά, σταθεροποίηση δηλαδή της ομαλικής κυβέρνησης και με την αποστολή κατάρτισης και εκπαίδευσης ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως σχεδιάζεται να γίνουν αυτές οι δράσεις στην Ουγκάντα ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε με κάποιες λεπτομέρειες πού βρισκόμαστε, ποιες χώρες είναι πρόθυμες να αποστείλουν ε, ανθρώπινο δυναμικό και τι γίνεται σε συνεργασία με τις ΗΠΑ βρίσκονται και στην ε, Ουγγάντα παρούσες για την ε, εκπαίδευση και κατάρτιση. Τι γίνεται σε ε, συνεργασία με τις ΙΠΑ από πλευράς μας, αν καταλήξουμε σε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Να επανέλθω σύντομα στη Βοσνία Εζεγοβίνη. Ο κύριος Βάγκελ ήδη έδωσε μια απάντηση. Δεν έθεσε ερώτημα, αλλά έδωσε μια απάντηση με την παρέμβασή του. Θα ήθελα να επανέλθω με μια απλή ερώτηση. Αναφέρθηκε ύπατος εκπρόσωπος σε σύνδεση με τις δυνάμεις μας εκεί. Υπάρχει μια άμεση διασύνδεση σε σχέση με εσά ή το συμβούλιο εφόσον θα υπάρχει ή το Συμβούλιο εφόσον θα υπάρχει παρουσία του, ε, της εκπροσώπου εκεί ή όχι. Ή το βλέπετε σε ανεξάρτητο πλαίσιο ύπατος εκπρόσωπο στη Βοσνία και ένοπλε δυνάμεις. Υπάρχει κάποια διασύνδεση ή όχι. Δεύτερη ερώτηση. Αναφέρατε την ε, Κίνα. Κίνα σε συνεργασία με το πρόγραμμα Αταλάντη. Υπάρχουν άλλα πεδία για τη συνεργασία με την Κίνα στο πεδίο, στο πεδίο της ασφάλειας ή το μόνο στοιχείο συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Κίνας σε θέματα ασφάλειας είναι αυτό. Συγκεκριμένα τώρα αναφέρομαι σε σχέση με τα θέματα ασφάλειας. Ευχαριστώ. Ζέμκε παρακαλώ. Jeśli można, to ja bym chciał tu nawiązać do dwóch kwestii, które mm, jak sądzę Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να πω ότι για τη δική μας ε, επιτροπή έχετε ιδιαίτερη σημασία εσείς ε, και ιδιαίτερα σε σχέση με τα όσα σας απασχολούν ε, κύριε Πρέσβη είναι πολύ ενδιαφέροντα για μας και για τις διεργασίες και τα συστήματα και τις, να δοκιμαστούν σε περιόδους κρίσης. Είχαμε δύο τέτοιες ε, καταστάσεις. Αφενός την καταστροφή των σεισμών στην ε, Αιτή που θα επανέλθω σε αυτό αμέσως και δεύτερον αυτό το οποίο έθιξε ο κύριος Πάσκου δηλαδή σε σχέση με την έκρηξη την ηφαιστειακή στο, στην Ισλανδία θα ξεκινήσω με το δεύτερο σημείο δηλαδή την Ισλανδία είχα την εντύπωση που αποκόμισα ότι μετά από αυτή την ηφαιστειακή έκρηξη υπήρξε μια χαοτική κατάσταση στην Ευρώπη και οι μόνοι που ενδιαφέρθηκαν να υπάρξει κάποια διέξοδος και το είπαν και ανοιχτά και ξεκάθαρα ήταν οι εταιρείε εναέριων μεταφορών διότι καθημερινά υφίστανται τεράστιες απώλειες από αυτή την κατάσταση. Τώρα, ερώτησή μου, σε κάποια τέτοια κατάσταση μπορεί να επανέλθουμε στο μέλλον. Ξέρουμε ότι η φύση, οι δυνάμεις της φύσης μας εκπλήσουν και μας ε, ε, πιάνουν πάντα εξαπίνης. Ε, λοιπόν, σε σχέση με το διεθνές πλαίσιο, για παράδειγμα, πέρα από τα κράτη-μέλη, τα τα κράτη. Υπάρχει δυνατότητα συντονισμένης δράσης ώστε να αντιδράσουμε συντονισμένα και οργανωμένα σε μια τέτοια κατάσταση διότι ξέρουμε ότι οι θεομηνίες και οι φυσικές ε, ε, καταστροφές δεν σταματούν στα εθνικά σύνορα, στα σύνορα μιας χώρας και γι' αυτό συμφωνώ σε σχέση με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Πάσκου. Πρέπει να πω ότι πραγματικά ανησυχώ ιδιαίτερα Ανησυχώ ιδιαίτερα βλέποντα ε, τι γίνεται σε σχέση με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που υιοθέτησαν μια πολύ παθητική, θα έλεγα αδρανή στάση. Και τώρα για την IT. Τώρα, σε σχέση με τις συζητήσεις, συζητήσεις των Υπουργών Άμυνας για παράδειγμα και, και σε σχέση και με την ε, Ισπανική Προεδρία υπήρξε προσπάθεια να συναχθούν κάποια συμπεράσματα από την έκδηλη αυτή κρίση στην ε, IT. Εγώ πιστεύω θα έλεγα ότι συμβαίνει το εξής ότι αυτή η φυσική καταστροφή με σαφέστατο τρόπο κατέδειξε ποια προβλήματα έχουμε στην Ευρώπη και πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το πρώτο πρόβλημα θεωρώ ότι ήταν το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε με υπερβολικά μεγάλη καθυστέρηση. Αυτό μπόρεσε κανείς να το δει και από τους τηλεοπτικούς σταθμούς ε, και από τις εκπομπές. Πιο γοργά και μια και βρίσκονται πιο κοντά αντέδρασαν οι ΙΠΑ. Αλλά είχα την εντύπωση πρέπει να πω ότι οι Ευρωπαίοι σε σχέση με την αντίδρασή τους ε, υπήρξε κάποια σύγχυση σε, σχέση με άλλες χώρες ε, δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε με ιδιαίτερα μεγάλη καθυστέρηση συγκρινόμενοι με άλλες χώρες. Και κάποιες ε, χώρες απέστειλαν ε, ομάδες ε, ε, διασωστών, αλλά όχι με συντονισμένο τρόπο. Και στο τέλος τι καταδείχθηκε, ότι τα ίδια τα ευρωπαϊκά μέσα παρέμβασης ήταν πάρα πολύ αποδυναμωμένα για τις εναέριες μεταφορές για παράδειγμα. Δεν έχουμε ούτε καν κοινό προϋπολογισμό για την κάλυψη τέτοιων δαπανών. Κύριε Πρέσβη, πολύ σωστά είπατε, πρέπει να συναχθούν τα συμπεράσματα από τέτοια μαθήματα. Ε, ποια μαθήματα είναι αυτά και ποια συμπεράσματα μπορούν να συναχθούν. Η κυρία Γκόμ Ευχαριστώ, ήταν πολύ καλή η παρουσία σας. Συμφωνώ και εγώ με τις ερωτήσεις των συναδελφών. Για την ενισχυμένη δομημένη συνεργασία. Και θα ήθελα να ρωτήσω εάν έχετε κάποιες πιο ε, συγκεκριμένε πληροφορίε ω προ τι προσπάθειε για το κράτο δικαίου. Ε, επιμένω κράτο δικαίου και όχι αστυνομία. Για το 2008 εμεί από το Κοινοβούλιο είχαμε επισημάνει ότι δεν έχει κανένα νόημα να γίνεται αυτή η τόσο καλή αστυνομική αποστολή εάν παράλληλα δεν γινόταν δουλειά και σε επίπεδο κράτου δικαίου. Και ναι, ανελήφθησαν κάποιε πρωτοβουλίε, αλλά ξέρουμε ότι δεν είχαν συνέχεια. επίσης για το Ιράκ θα ήθελα να ρωτήσω και ξέρω ότι έγινε και μια πρώτη συνεδρίαση σε σχέση με τα όσα έχετε σημειώσει στο Ιράκ και με προοπτική το 2012. Ασφαλώς είναι πολύ ε, ενδιαφέρουσα και σημαντική η αποστολή, αλλά λειτουργεί υπό την καθοδήγηση του Βρετανικού σκέλους. Έχει δηλαδή τους περιορισμούς τους Βρετανικούς σε σχέση με την ασφάλεια και την άμυνα γιατί εμείς από το Κοινοβούλιο είχαμε ζητήσει να αυτονομηθεί η ευρωπαϊκή παρουσία. Ξέρω ότι παραχωρήθηκαν κάποιοι χώροι στην ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία εκεί, κάποιες εγκαταστάσεις. Ε, έγινε όντως αυτό και διευκόλυνε σε τίποτε. Για τη Σομαλία, με λύπη μου σας λέω ότι από αυτά που μας είπατε, από αυτά που γνωρίζουμε, από αυτά που διαβάζουμε, δυστυχώς δεν έχω πιστεί ως προς την ε, σκοπιμότητα, αποτελεσματικότητα αυτής της ε, αποστολής. Δεν είμαστε καθόλου πεπισμένοι ότι δεν θα καταλήξουν αυτοί που εκπαιδεύουμε στην υπηρεσία της Χασαμπάπ. Ξέρω ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, αλλά είναι πολύ επικίνδυνο αυτό το παιχνίδι. Κόγκο. από αυτά που βλέπω στην έκθεση, πιστεύω ότι δεν κάνουμε και τίποτα διαφορετικό. Δεν αλλάζουμε τίποτε δηλαδή. Δεν δίνουμε απαντήσεις στο ζήτημα της ε, ε, πάταξης των πολύ σοβαρών ε, προβλημάτων παραβιάσεων των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών, δηλαδή σεξουαλική εγκληματικότητα που υπάρχει εις βάρος τους. Όταν δεν αναλαμβάνουμε δράση σε αυτό το φοβερό πράγμα σε αυτή την κατάφορη παραβίαση των πρώτων δικαιωμάτων, τι κάνουμε στο Κονγκό. Δεν ήρθε η ώρα πια να το ξαναδεί το Συμβούλιο αυτό, το θέμα του Κονγκό, την αποστολή και να φροντίσει να υπάρχει επαρκές, προσωπικό επαρκής δυνάμεις καλύτερα, με επαρκή εντολή για να απαντήσουν τα προβλήματα. Το ίδιο θα μπορούσατε να σας πω και τη Γουινέα Μπισάου. Δηλαδή, όταν μπορούμε να προσφέρουμε κάτι. Μην, μιλάμε, μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για χώρα η οποία ε, είναι πολύ σημαντική για μας. Ε, έχουμε πολιτικές εξελίξεις οι οποίες θα έπρεπε κανονικά ε, να μην έχουν συμβεί. Δηλαδή αν είχε η αποστολή μας κάποια αποτελέσματα δεν θα έπρεπε να ήταν αυτές οι πολιτικές εξελίξεις. Άρα, πού πάμε και τι κάνουμε και γιατί, να, γιατί είναι η κατάσταση αυτή. Θα προτιμούσα βέβαια να παραμένουμε εκεί, αλλά με, τη σωστή, με το σωστό δυναμικό, με τη σωστή μέθοδο, έτσι ώστε να φέρουμε αποτελέσματα, πράγμα που δεν φαίνεται να συμβαίνει. Επίσης, ως προς, τον, ως προς την υπηρεσία, έχουμε καταφέρει πια να έχουμε πολυετή προϋπολογισμό, αυτόν ακριβώς τον οποίο είχαν αποτρέψει, είχαν, στον οποίο είχαν θέσει τόσα προσκόμματα οι Βρετανοί φίλοι. Καταφέραμε να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια. Η κυρία η Λέιδη Άστον ε, επέφερε κάποια αλλαγή. στην τελευταία ανάλυση Βρετανίδα. Είναι, είναι και επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικών ε, σχέσεων της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλισης εν ολίγης. Και εν τέλει, έχουμε τεράστια και ανευπροηγουμένου οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Όλοι είμαστε στρατιωτικοί στις χώρες μας πιέζονται, έχουν μεγάλο, υφίσταται πολλές πιέσεις και άγχος, περικοπές από το προπολογισμό τον εθνικό, από τους εθνικούς προπολογισμούς. Οι υπουργοί τα συζήτησαν όλα αυτά. Σε ποιο βαθμό επηρεάζονται οι ικανότητες που είχαμε πει ότι είναι απαραίτητες και ελάχιστες για τις αποστολές, δηλαδή τελικόπτερα. Και όταν είναι η συμφωνία στον τομέα αυτών ε, επιτοπλίστων ε, σπηλωμένες από βρώμικες συμβάσεις και δεν όχι μόνο στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα, με τη Γαλλία, τη Γερμανία και τα λοιπά, τα υποβρύχια. Πώς θα μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε την εικόνα. Ευχαριστώ κύριο Κυρίλοφ παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Πρεσβευτά. διάβασα μια έκθεση πρόσφατα και γι' αυτό αποφάσισα να θίξω το ζήτημα, γιατί δεν άκουσα να γίνεται κουβέντα πουθενά για τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Και θυμάμαι ότι ούτε για την Νότια Οσετία και την Απχασία ακούγαμε τίποτα. Μέχρι που ξαφνικά ξεσπάσανε τα πάντα και ανακαλύψαμε ότι υπήρχαν προβλήματα για τα οποία κανεί δεν μα είχε μιλήσει. Στον Ακόρνο Καραμπάχ, λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι, από τι τελευταίε εκθέσει που έχω παρακολουθήσει, είναι ο απερχόμενος συμπρόεδρος της ομάδας του Μίνσκ, ο Ρώσος, και ο νέος συμπρόεδρος, πάλι, της ομάδας του Μίνσκ, πάλι Ρώσος, μαζί με τον Αμερικανό πήγαν στο Αζερβαϊτζάν, συζήτησαν τον πρόεδρο εκεί, συζήτησαν, ε, ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, μια δυναμική αναπτύσσεται, ελπίζω να μας βγει σε καλό, για την ρύθμιση, για τη διευθέτηση αυτής της σύγκρουσης. Και φαίνεται ότι συμφωνήθηκε και μάλιστα έγινε και κοινή δήλωση με την έγκριση του Γάλλου Συμπροεδρού και από την ομάδα εργασίας για τον Κάφκασο έλαβα πολύ σημαντική υποστήριξη πρέπει να σας πω για τη σύσταση που μας επιτρέπει τώρα μετά την συνθήκη της Λισαβόνας να, η συνθήκη της Λισαβόνας να μάλλον τα θέση σε ισχύ να αναλάβουμε την πρωτοβουλία. Και γιατί θέτω το ερώτημα, διότι δεν μιλήσατε καθόλου για τη σύγκρουση στο ε, Ναγκόρνο Καραμπάχ. Με κάποιο τρόπο, από ό,τι φαίνεται όμως, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει. Και για απεμπλοκή, εάν υπάρξει απεμπλοκή, η ειρηνευτική πρωτοβουλία και δραστηριότητα δεν βλέπω ποιο μπορεί να διαδραματίσει με πιο πιστικό τρόπο από ότι εμεί, γιατί άλλοι ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι, η Ρωσία και οι Αμερικανοί. Δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει δράση. Δεν θα αρχίσουμε να συζητάμε λοιπόν ή θα περιμένουμε πρώτα να γίνει κάτι και μετά να αρχίσουμε να το συζητάμε. Ευχαριστώ κύριε Πρεσβευτά. Ο γύρος του κόσμου. Σε 8 δευτερόλεπτα. Ίσως μπορείτε να παρουσιάσετε τις απαντήσεις σας σε ομάδες, γιατί είναι αρκετά κοινά τα θέματα. 80 ημέρες, δεν είπαμε, λέει ο Πρόεδρος. Έχετε μισή ωρίτσα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ όλους όσοι έθεσαν ερωτήσεις και διατύπωσαν παρατηρήσεις. Με χαρά βλέπω ότι ε, προκαλεί τέτοιο ενδιαφέρον και γεννά τόσο ερωτηματικά η παρέμβασή μου. Και στα αγγλικά θα έλεγα ότι τίνω να συμφωνήσω, ο κύριος Γουακέ δεν είναι εδώ, με τον κύριο Γουατιέρη, τίνω να συμφωνήσω όταν κάνει τις σχετικές ερωτήσεις και με την κυρία Γκόμες όμως, γιατί έχετε τα ίδια, σας απασχολούν τα ίδια ερωτηματικά που απασχολούν και εμένα σε ορισμένε περιπτώσεις, χωρίς δυστυχώ να έχω πιο πολλές απαντήσεις από ότι εσεί για τα θέματα που σα απασχολούν. Θα προσπαθήσω όμως να τα εκθέσω με ένα συστηματικό τρόπο, ξεκινώντας από τα θεσμικά. Κάποιος εξημών ρώτησε για την μόνιμη δομή, για τη συνεργασία μάλλον της μόνιμη δομής. Και γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω από τον κύριο Γκάλερ και την κυρία Γκόμες που έθιξαν το ερώτημα. <clears throat> Πιστεύω πως είναι ένα θέμα που κάποιοι ρώτησαν αν συζητήθηκε στο δείπνο των Υπουργών να μείνεις πολύ πολύ σύντομα. Μόνο ένας υπουργό, ο υπουργό ε, θα πούν η Υπουργό Τσακών, η Ισπανίδα ε, Υπουργό, είπε ότι έγινε ένα σεμινάριο. Ποιο ήταν τα αποτελέσματα, ήταν ένα είδος brainstorming, να προσπαθήσουν να βρουν ιδέε κτλ. Η ιδέα ήταν αν αυτή η δομή η μόνιμη συνεργασία υπήρχε ήδη ή όχι. Και ορισμένοι λένε πω ναι, υπάρχει γιατί Δεν είναι η ιδέα του EDA, δεν είναι η ιδέα των ομάδων ε, μάχης. Ε, κάποιοι ρώτησαν αν υπάρχουν μία ή δύο ή περισσότερες δομές. Εμείς κάνουμε μία μόνιμη δομή συνεργασίας και περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξουμε. Ξέραμε πολύ λίγα πράγματα όταν άρχισε να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας και το πρωτόκολλο που λέει ότι πρέπει να μην είναι... να υπάρχει βούληση και συνεργασία για να μπορέσει να προχωρήσει ο τομέας αλλά και να υπάρχουν τα βιομηχανικά, τα και τεχνικά μέσα, ώστε κάποιες από τις χώρες να προχωρήσουν. Αυτού του είδους οι ομάδες υπάρχουν. Είναι ένα από τα πιο ανοιχτά ζητήματα μέχρι στιγμής όσον αφορά την ε, εξέλιξη της συνθήκης της Λισαβόνας. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι όπως και πολλά άλλα στη συνθήκη της Λισαβόνας. Μία από αυτές τις ιδέες που ήρθαν από το προηγούμενο σχέδιο κειμένου του συντάγματος που δεν υπήρξε ποτέ, ήρθαν στην συνθήκη της Λισαβόνας, ενώ εντωμεταξύ έχουν γίνει διάφορα πράγματα. Άρα λοιπόν έχουμε κάποια στοιχεία που μπορεί να θεωρηθούν τμήμα αυτής της ε, μόνιμης δομής συνεργασίας. Έχει γίνει λοιπόν ήδη κάποια δουλειά από αυτόν. Για τον ε, θεσμικό τομέα με ρωτήσατε για την, υπηρεσία, την εξωτερική υπηρεσία και υπήρξαν κάποια ερωτήματα τα οποία δεν έχουν ακόμα επιληθεί και που είναι εξαιρετικά σημαντικά και που θα πρέπει να λυθούν. Κύριος αφορούν τις σχέσεις νομίζω ο κύριος Πάσκου το ρώτησε αυτό και ο κύριος Γκάλερ και άλλοι και ο κύριος Ζέμκο με ρώτησε για το ίδιο πράγμα. Τη σχέση μεταξύ του CMPD και το είπα του εκπροσώπου. Αν υπάρχει άμεση ή έμεση σχέση. Και επίσης η διαφορά ανάμεσα στα δύο οργανογράμματα το οργανόγραμμα Μπροκ και και το οργανόγραμμα του Συμβουλίου, τα οργανογράμματα είναι οργανογράμματα. Για μένα δεν είναι και τόσο σημαντικά, γιατί αυτό που κάνουν από την εμπειρία μου είναι κάτι το κινούμενο. Ε, προσπαθείς να φτιάξεις ένα σπίτι, φτιάχνεις ένα σχέδιο και όταν έχεις θέσει τα μισά της οικοδομής, θυμάσαι πως ξέχασες να βάλεις τα μπάνια και πρέπει να αλλάξεις τα σχέδια ή την ηλεκτρική εγκατάσταση. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ένα βασικό σχέδιο για το τι θέλεις να πετύχεις και αυτό είναι το οργανόγραμμα. Αλλά δεν υπάρχουν στο οργανόγραμμα αυτές οι μικρές γραμμές που συνδέουν τις διάφορες ε, ε, υπηρεσίες. Δηλαδή η αλυσίδα Ενημέρωση. Οι στρατιωτική είναι πολύ καλοί, βάζουν διάφορα χρωματάκια, ε, διάφορα συνδέονται με μπλε, ε, άλλα με, κόκκινο, με κίτρινο, σαν να είναι καλώδια που συνδέουν τα οργανόγραμμα και λέει ποιο δίνει τις διαταγέ σε ποιον, ποιο συντονίζει ποιον και σε ποιον πρέπει κανεί να αναφερθεί. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα. Και το να πιστεύουμε ότι το CMPD θα αναφέρεται μόνο στον ύπατο εκπρόσωπο, ίσως να γίνει έτσι. Αλλά είναι, δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό, γιατί ο ύπατος εκπρόσωπος θα καταξιδεύει πολύ και το CMPD θα πρέπει καθημερινά να λαμβάνει αποφάσεις και μάλιστα άρθμες αποφάσεις καθημερινά. Οπότε χρειάζεται ένα δεύτερο επίπεδο ό,τι και να αποκαλέσουμε το ενδιάμεσο επίπεδο, θα υπάρχει μια σύνδεση και μια ανάγκη οργάνωσης. Τελευταία, έχω χάσει τον μπούσουλα. Όπως και εσείς, περιμένω και εξαρτάμαι από το τι μας πει ο κύριος Κριστόφερσεν. Η Κορεπέρ είναι πολύ πιο καλά ενημερωμένη για την υπηρεσία εξωτερικών ε, δράσεων. Αυτό το κάνουν, ε, ασχολούνται με αυτό καθημερινά. Πιστεύω ότι υπάρχουν δύο συστήματα. Ένας από τους δύο γενικούς γραμματείς ή τους τρεις γενικούς γραμματείς, ένας από αυτούς είναι πιο διαχειριστής, ο ένας είναι διαχειριστής, ο άλλος είναι πολιτικός ε, διαχειριστής και ο άλλος δεν ξέρω εγώ τι. Πάντως θα υπάρχει σύνδεση σε κάθε περίπτωση μέσω αυτού του δευτέρου επίπεδου. Υπάρχει λοιπόν άμεση σύνδεση της διαχείρισης κρίσεων με το ανώτερο επίπεδο. και ούτω καθεξής. Ε, θα υπάρχει μια σύνδεση κατακόρυφα προς την κορυφή του Ολύμπου, αν θέλετε να το πείτε και έτσι. Δεύτερο. Και στη συνέχεια, ίσως για να ολοκληρώσουμε κιόλας, σε σχέση με ερωτήσεις, ερωτήματα που συσχετίζονται με θεσμικές πτυχές, θεσμικά ζητήματα. Ναι, ήταν αυτές οι δύο τελευταίες ερωτήσεις της κυρίας Γκόμες για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας και την αντιμετώπιση κρίσης. Ξέρετε, υπάρχουν πολιτή προγράμματα σε σχέση με την υπηρεσία άμυνα. Υπάρχει και το θέμα έγκριση όμω εδώ, το οποίο πολλέ φορέ εγκρεμεί Η κυρία Άστον δεν είναι μέλο τη Βρετανική κυβέρνηση, δεν έχει ψήφο λοιπόν. Και παρότι Πιστεύω ότι νομίζει και θεωρεί η κυρία Άστον ότι ένα τέτοιο πολιετές ε, πρόγραμμα θα ήταν πολύ καλύτερο για το έργο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας. Δεν έχει λέγει, δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει. Αν, για παράδειγμα, κάποιος, ε, κάποια κυβέρνηση πει όχι. Και ήμουν εγώ παρόν όταν είπε ο Βρετανός ε, υπουργό ότι δεν θα δεχόταν κάτι τέτοιο, άρα δεν θα μπορούσε να προχωρήσει. Παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο, δεν ακούγεται three days elections. Σε τρεις μέρες θα έχουν εκλογές εκεί, ναι, εντάξει. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε το τι θα γίνει ακριβώς. Όμως η κρίση, η κρίση είναι σημαντικό πράγμα, διότι έχει επιπτώσεις στο έργο της ε, EDA, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας, Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άνημινας και για την έκθεση του Αλεξάνδρε Βάης στους υπουργούς επέμεινε και ενέμεινε ότι πρέπει να μάθουμε κάτι και να υπάρξει κάποια ε, εξοικονόμηση ε, όσον αφορά και τη συνεκτικότητα των δράσεων και των προγραμμάτων. Θα μπορέσουν να εξοικονομηθούν κονδύλια. Ανέφερε για παράδειγμα το θέμα του προγράμματος Eurofighter του ε, Ευρωπαϊκού Πολεμικού Καταδιοκτικού Αεροπλάνου με χώρες που συμμετέχουν στο εγχείρημα αυτό και υπάρχει και ένας ανταγωνισμός, μια ανταγωνιστική σχέση σε σχέση με το Γαφάλ, το γαλλικό πολεμικό αεροπλάνο, σε σχέση για παράδειγμα με τα όσα επενδύουν οι Αμερικανοί σε σχέση με την εξέλιξη ενός ε, και μόνου πολεμικού αεροπλάνου. Υπάρχει λοιπόν θα έλεγα πολυσχηδής προσπάθεια από πλευράς μας ε, αλλά περί αυτού πρόκειται για την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και για τις δράσεις ε, ή τα, τις δραστηριότητες ε, αλλού στον κόσμο. Βοσνία Ζεγοβίνη εκφράστηκε μεγάλο ενδιαφέρον. Πρώτον, ο κύριος Πάσκου ανέφερε για την εκπαίδευση. Σίγουρα, ναι, γίνεται αυτό και ποια είναι η ε, non-executive ε, αποστολή για να ε, όχι μόνο εποπτεύουμε αλλά και για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε. Είναι μια νέα γενιά αυτή, έχετε δίκιο, πρέπει να την εκπαιδεύσουμε και να οδηγηθεί σε κατάρτιση. Και μια νέα γενιά βρίσκεται ήδη εκεί και αλλάζουν τα πράγματα επιτόπου και αυτό είναι καλό, καλά μαντάτα. Τα περισσότερα καλά μαντάτα που έχουμε σε σχέση με τη Βοσνία Ζεγοβίνη προέρχονται από τους στρατιωτικούς και όχι τόσο στο πολιτικό επίπεδο. Μετά κάποιοι για την αξιολόγηση κινδύνου και κινδύνων και την ανάγκη που τόνισε ο κύριος Βάγκερ για τι βρισκόμαστε εκεί, τι κάνουμε και ποιοι είναι οι στόχοι μας και ότι πώς χρησιμοποιούμε τις δυνάμεις μας εκεί επί τόπου. Τώρα για τις ένοπλες δυνάμεις που βρίσκονται στη Βοσνία χίλιοι περίπου σε τρεις ομάδες ή σε τρεις κατηγορίες ε, δράσεων. Η μία είναι η ανάγκη να είμαστε παρόντες εκεί. Επιμελητιακή υποστήριξη, παροχή ε, εξυπηρέτησης, ε, επιμελητιακή κτλ. όταν βρισκόμαστε επί τόπου. Το δεύτερο, δεύτερη κατηγορία. Οι ένοπλες δυνάμεις οι οποίοι ασχολούνται με ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ε, από όλη την επικράτεια σε σχέση με την επικράτεια της Βοσνίας Εζεγοβίνης, ώστε να ειδοποιούμαστε έγκαιρα αν υπάρχει κάτι στραβά. Το θέμα ή το ερώτημα δεν είναι μόνο σε σχέση με μια αντιπαράθεση μεταξύ ε, εθνοτικών κοινοτήτων ή ανταρτών, ανταρτικών μονάδων, αλλά για παράδειγμα κάποιου μεμονωμένου συμβάντος ή γεγονότος κάποιας εκτροπής κάποιες εβδομάδες πριν από τις εκλογές αν κάτι είχε συμβεί σε ένα μικρό χωριό για παράδειγμα. Ίσως ακόμα και ένα αυτοκίνητο που χτυπάει κάποιο πεζό, ένα νέο ή μια γυναίκα που πάει να περάσει ένα δρόμο και είναι οδηγός από μια διαφορετική κοινότητα σε σχέση με εκείνον που έχει πληγωθεί, έχει τραυματιστεί, έχει σκοτωθεί, παίρνει διαστάσει αυτό. Και όλα αυτά μπορούν να προληφθούν στις διαστάσεις που μπορούν να πάρουν μετά ανεκράγει να υπάρχει μια εκρυθμή κατάσταση. Αυτού του είδου τα πράγματα που μπορούν δηλαδή να προκαλέσουν μεγάλη βία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν χρειάζονται πάρα πολύ ένοπλοι γι' αυτό, αλλά πρέπει να υπάρχει εποπτεία και πρόληψη, να υπάρχει εκτελεστική αρμοδιότητα και εξουσία, να μπορούμε να είμαστε εκεί παρόντες με παράδειγμα κάμποσους, κά, κά, κάποιες δεκάδες ένοπλους ώστε να σταματήσει η έκρηθμη βία σε ένα χωριό εκεί και φυσικά από κοινού σε συνεργασία με τους Βόσνιους να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τα πράγματα και να μην υπάρξει μια διάδοση, ας το πω έτσι, της φωτιάς και πάρει διαστάσεις το πρόβλημα. Παράδειγμα, όταν υπάρχουν προβλήματα ταυτόχρονα σε κάποια χωριά και που μπορούν να δημιουργήσουν μια ανάφλεξη, αν δεν δράσουμε έγκαιρα δεν θα μπορέσουν να, να αντιμετωπιστούν αυτά από την αρθία ή από μεγαλύτερες ένοπλες ε, δυνάμεις. Πρέπει να γνωρίζουμε λοιπόν ότι υπάρχει ανάγκη για να είμαστε παρόντες και να προλαμβάνουμε τα πράγματα πέρα από την επιμελητιακή παρουσία χρειαζόμαστε εκτελεστική παρουσία ώστε άμυνα να υπάρχουν οι ένοπλες δυνάμεις που θα μπορούν να αποσταλούν έγκαιρα για να σταματήσει η έκρηθμη βία και οι, ε, οι βιοπραγίες έγκαιρα όπου παρουσιάζονται. Αυτά σε σχέση τώρα με την ε, Βοσνία και το σκηνικό το σενάριο εκεί. Δεύτερο θέμα το οποίο και αυτό ενδιέφερε πολύ και πηχήθηκε στις παρεμβάσεις ήταν η Σομαλία και η κατάρτιση εκπαίδευση στην ε, Ουγκάντα για αυτές τις δυνάμεις. Για την εκπαίδευση ο κύριος Γκάλερ ρώτησε για τη συνεργασία με τις ΗΠΑ. Ναι, υπάρχει συνεργασία με τις ΗΠΑ, διότι παρέχουν τις μεταφορικές δυνατότητες ε, ώστε αυτοί οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να πηγαίνουν εκεί να μεταφέρονται εκεί, δίνουν επίσης και κονδύλια παρέχουν και είναι σε επαφή και υποστηρίζουν την κυβέρνηση της ε, Ουγκάντα για να μπορέσουν ε, αυτά τα επιτελεία σε ένα αρχηγείο, ας το πω έτσι, να συνταθούν στην Καμπάλα, στην πρωτεύουσα της Ουγγάντα. Και είναι και το θέμα της ε, υποστήριξης με κονδύλια. Τώρα, σε σχέση με αυτό το οποίο είπατε κυρία Γκόμες για την επιστροφή στην Άσαμπα. Έχουμε τις ίδιες εγγυήσεις που δίνονται όταν εκπαιδεύουμε για παράδειγμα Αφγανούς αστυνομικούς, όταν το ΝΑΤΟ εκπαιδεύει τέτοιες δυνάμεις σε σχέση με την ε, επέμβαση σε συγκεκριμένες περιοχές. Όταν και εμείς εκπαιδεύουμε κάποιους αστυνομικούς και μετά κάποιοι οδηγούνται σε κάποια έκτροπα. Δεν, είναι, δεν υπάρχει εγγύηση ότι όλοι όσοι θα εκπαιδεύονται από εμά θα είναι πάντα υποδείγματα στη συμπεριφορά τους και δεν θα εκτραπούν ποτέ. Είναι πολύ πιο δύσκολο, ακόμα πιο δύσκολο σε χώρες που βρίσκονται σε ένοπλη σύραξη. Όμως και η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι απρόβλεπτη. Εκείνο το οποίο μπορεί να προβλέψει κανείς είναι τουλάχιστον η αναγκαία σωστή κατάρτιση και εκπαίδευση ώστε να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε, να δημιουργήσουμε τέτοια άτομα που θα είναι καταρτισμένα να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. 100% βεβαιότητα δεν είναι ε, διασφαλισμένοι ποτέ και δεν είναι δυνατόν εφόσον δεν είναι διασφαλισμένη αυτή η 100% πρόβλεψη να μένουμε εμείς αδρανείς. Και τώρα για τη Σομαλία και το θέμα της δράσης Αταλάντη. Νομίζω ότι ο κύριος Γουαλτιέρη ήταν εκείνος που μας, με ρώτησε αν αυτό το οποίο συνέβη στην μεταξύ Μάρ και Ασσαμπά. αυτές είναι ε, ομάδες φιλάρχων, στρατιωτικές ομάδες ε, πολεμάρχων και φιλάρχων που βρίσκονται σε ανταγωνισμό και σε σύγκρουση. Δεν είναι το θέμα της δημιουργίας ενός νέου κράτους, αλλά το να αποκτήσουν εξουσία και να ελέγχουν εκείνη τα πράγματα στην περιοχή τους. Η βάση εκείνη που κατέλαβαν και σε σχέση με τις, ε, τα έσοδα από την πειρατεία που ε, τους κάνουν να θέλουν να ελέγχουν αυτή την περιοχή με αυτή τη βάση και αυτές τις δράσεις. Αυτοί οι νέοι, αυτές οι ομάδες ε, αγόραζαν αυτοκίνητα, όπλα, έχτιζαν, δαπανούσαν κονδύλια, όλα αυτά είναι, ας το πω έτσι, ένα κίνητρο για να μπορούν να, να κινητοποιούνται αυτοί, να, να πηγαίνουν και να δρουν με αυτόν τον τρόπο εκεί. Αν με ρωτήσετε όμως και θέσετε το ερώτημα κυρία Γκόμες πότε θα σταματήσει αυτό κάνοντας εμείς, ακολουθώντας αυτές τις δράσεις ε, και αναφέρθηκε πιο πριν ότι υπάρχει η καταδίωξη, αν υπάρχει καταδίωξη λέμβων, πειρατικών λέμβων στο ανοιχτό πέλαγος. Εμείς προσπαθούμε να διασφαλίσουμε το πλαίσιο ασφάλειας, να δημιουργήσουμε ασφάλεια όσον αφορά τα πλοία μας που κυκλοφορούν και ε, διέρχονται από αυτή την περιοχή, η θαλάσσια περιοχή. Δεν είναι όμως το θέμα μόνο το θέμα πλοίων. Χρειαζόμαστε και αεροπλάνα και ελικόπτερα Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η πειρατεία δεν θα είναι πια κίνδυνος και απειλή και κερδοφόρα δραστηριότητα εκεί και πρέπει γι' αυτό να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα. Την ίδια την κατάσταση στη στεριά, στην ξηρά και όλο τον ε, κύκλο της ε, ε, της αλυσίδας του χρήματος και της ροής του χρήματος και το πώς μπορεί ε, να αντιμετωπιστεί αυτός ο κύκλος της κερδοφορίας, της πειρατείας. Αυτό είναι θέμα του οποίου έχει επιληφθεί η Πολιτική και Στρατιωτική Επιτροπή για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα στη Σομαλία. Και μετά μου τέθηκε το ερώτημα, ναι, κάποιες ερωτήσεις ε, για τον Νότιο Κάυκασο υπήρξε μέλος που εξέφρασε ενδιαφέρον να πληροφορηθεί για το τι τεκταίνεται εκεί και επίσης ε, ένα ερώτημα για το πρόβλημα, το ζήτημα του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Το Ναγκόρνο Καραμπάχ είναι το πιο ε, εύκολο αν θέλετε να απαντηθεί μια και δεν έχουμε αποστολή εμείς δεν υπάρχει κάτι να εκθέσω για το τι κάνουμε σχετικά εκεί αυτό όμως που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε και να είμαστε σε επαφή ώστε να διαμεσολαβήσουμε και να δώσουμε πολιτική και διπλωματική υποστήριξη. Η κατάσταση στον Αγκόνο Καραμπάχ εντωμεταξύ υπήρχε, υπήρχαν κάποιες ελπίδες πριν από έξι μήνες, αλλά μια και οι Αρμένοι είχαν την, το θέμα της ε, επαιτίου που εορτάστηκε τα πράγματα πήγαν στραβά σε σχέση με τις σχέσεις με την Τουρκία, μεταξύ Αρμενίας Τουρκίας και τώρα δεν ξέρουμε αν η συμφωνία που είχε ε, συναυθεί αν θα μπορέσει να υλοποιηθεί και να εφαρμοστεί ή όχι μεταξύ Αρμενίας και Τουρκίας. Αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα. Τώρα αν η ΕΕ θα είναι εκείνη που θα πρέπει να επιλύσει το πρόβλημα αμφιβάλλω αν θα μπορέσει να γίνει αυτό, αλλά θα έχει ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό είναι το θέμα τώρα. Μέσα στην, ε, στο πλαίσιο της ε, ε, ευρωπαϊκής πολιτικής όλες οι χώρες αυτές η Τουρκία, η Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν και η, Αρμενία μέσα στο πλαίσιο της εύξηνης συνεργασίας, της συνεργασίας στον εύξηνο πόντο στον Κάφκασο θα πρέπει να μπορούν να είναι σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορούμε να συνεισφέρουμε για την επίλυση. Τώρα για την Απχαζία, Απχαζία και την ε, ε, Νότια Οσετία για το πρόβλημα το οποίο εθίγει από τον ε, από το μέλος δεν βλέπω στρατιωτικές δυνάμεις, σίγουρα όχι στην Απχαζία ή στην Νότια Οσετία με τους Ρώσους, από κοινού με τους Ρώσους. Δεν ξέρω αν κατανόησα και απόλυτα καλά το ερώτημά σας. Τώρα, για παρατηρητές ε, που θα μπορούσαν να αποσταλούν σε αυτές τις περιοχές, ε, διότι αποδεικνύεται ότι είναι μια πολύ σημαντική αποστολή η UMN, η μόνη που είναι παρούσα στη Γεωργία από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωση που οδηγεί τα πράγματα σε κάποια κινητοποίηση και για την ε, δυνατότητα να, να περνούν τα σύνορα από την Νότια Οσετία προς την Απχασία. Αρχίζουμε να και εργαζόμαστε από κοινού με το, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε τον ε, Γενικό Γραμματέα. Ο Γενικός Γραμματέας ε, διόρισε ένα νέο ειδικό απεσταλμένο για αυτό το ζήτημα. Είχα ένα γεύμα μαζί του την προηγούμενη Παρασκευή και συζητήσαμε και αυτό που συμβαίνει είναι να δούμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί, να ληφθούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, να μπορέσουν οι δύο κοινότητες ε, ένθεν και ένθεν των συνέρων να, των συνόρων με συγχωρείτε, να βελτιώσουν την, ε, το θέμα εμπιστοσύνης, να οικοδομήσουν ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ τους, οικονομικές συναλλαγές, ε, λοιπά. Θα πρέπει να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να προωθήσουμε την ιδέα του Υπουργού για Μποκασβίλη, για παράδειγμα, σε σχέση με αυτή την πρωτοβουλία ενσωμάτωσης, ε, ολοκλήρωσης περιφερειακής μεταξύ Οσετίας και Απχασίας. Πρέπει να βρεθούν οι όροι για αυτή την πρόταση, ιδιαίτερα σε ένα νομικό, στην αποσαφήνιση των νομικών όρων θα πρέπει να ε, εργαστούμε περισσότερο για τα μέτρα οικοδόμησης ε, εμπιστοσύνης. Αναφερθήκατε εσείς ε, στη διαδικασία της Γενέβης για τη Γεωργία. Η διεργασία αυτή έχει κάτι το θετικό σχετικά. Είναι μια παγιωμένη μετά από τις διαβουλεύσεις και συζητήσεις, είναι τώρα μια μια διαδικασία που έχει παγιωθεί. Υπάρχουν συναντήσεις τώρα σε τακτά διαστήματα. Μετά από τη δεύτερη συνάντηση είχε αναφερθεί, θα είναι η δεύτερη είχα πει και θα είναι μάλλον η τελευταία. Λάθος είχε γίνει, δεν ήταν η τελευταία. Τα πράγματα κινούνται με αργούς ρυθμούς, αλλά προχωρούν. Και αυτό είναι το καλύτερο σε σχέση με αυτό. Αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι θέλουν να είναι παρόντες και να, είναι, να εκπροσωπούνται εκεί, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να διαβουλεύονται και να συζητούν και να προχωρούν τα πράγματα. Ακόμα και αν δεν υπάρχει μεγάλη πρόοδος και δεν κινητοποιούνται γοργά τα πράγματα και δεν επιλύονται πιο γοργά υπό πρακτικούς όρους. Αυτό σε σχέση με την ενημέρωσή σας, ε, εν συντομία, τώρα κάποια πράγματα πολύ σύντομα, σύντομα ε, για την ε, Κίνα. Γνωρίζω ότι σε σχέση με το ε, υπουργικό επίπεδο είχε επιστρέψει η κυρία Άστον όσον αφορά την ε, Σανγκάη έχει συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να μπορούμε να συζητούμε με τους Κινέζους. Η Αταλάντη είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα, διότι 90% του εμπορίου Κίνας-Ευρώπης περνά από αυτή την ε, ζώνη, από αυτή την περιοχή. Πρέπει να βρούμε λοιπόν κομβικά σημεία που θα υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον για να συζητούμε και να διαβουλευόμαστε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, για παράδειγμα, με τους ε, Κινέζους είναι δύσκολο να μπορέσουμε να κινηθούμε. Έχουν τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας οι Κινέζοι σε σχέση με εμάς. Αλλά σε κοινά σημεία τα οποία μας απασχολούν κομβικού χαρακτήρα θα μπορούσαμε να έχουμε διαβουλεύσεις για τα θέματα ασφάλειας με τους Κινέζους. Τώρα για το θέμα και του Ιράκ. ξέρετε ότι η ασφάλεια είναι το μεγαλύτερο θέμα στο ε, ε, Έχουμε παρουσία εκεί από την Βαγδάτη δεν έχουμε ακόμα μετακινηθεί ε, εκτός ε, της ε, Βρετανικής περιοχής. Το θέμα της δαπάνης και διάθεσης κονδυλίων για αυτή την αποστολή είναι ζωτικού χαρακτήρα. Όμως προς το παρόν είμαστε ασφαλείς, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε όσον αφορά το κτίριο το βρετανικό, αλλά θα μετακινηθούμε στο βόρειο τμήμα στο βόρειο τμήμα του Ιρακ. Θα προσπαθήσουμε να πάμε και στην Πάσρα αν είναι δυνατόν για να καταφέρουμε να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να επεκτείνουμε το πεδίο. Για το Κονγκό και στην ε, ε, ΚΕΠΑ θα πρέπει να δούμε ακριβώς ε, σε λεπτομέρεια το τι είναι αυτό το οποίο κάνουμε στο Κονγκό. Το ίδιο ισχύει και για την Γινέα Μπισάου για την αποστολή. Η αποστολή απέτυχε σε σχέση με τον, την διασφάλιση του τομέα της διαφύλαξης της ασφάλειας σε σχέση με τους ναρκοεμπόρους που έχουν την εξουσία και που κάνουν εκεί κουμάντο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτοί είναι εκείνοι που βρίσκονται στην εξουσία αυτή τη στιγμή και απέτυχε η δράση μας. Για το ηφαίστειο και πάλι δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια όλων. Η διαφορά τώρα μεταξύ σεισμού και ε, ηφαιστείου, ο σεισμός προκάλεσε ανθρωπιστική ε, καταστροφή. Η ε, έκρηξη του ηφαιστείου δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα σε εταιρείε εναέριων μεταφορών και σε προβλήματα που είχαν ταξιδιώτες ε, στην Ήπειρο της Ευρώπης το τι μπορούμε να μάθουμε σε σχέση με την ε, ηφαιστειακή έκρηξη. Ε, εγώ ίδιος είχα ξεμείνει ε, στις Βρυξέλλες, δεν μπόρεσα να πάω στη Μαδρίτη, είχα συνάντηση εκεί και πάλι όμως χιλιάδες, μιλιάδες, εκατομμύρια πολίτες έχασαν την δυνατότητα να μετακινηθούν, δεν μπορούσαν να μετακινηθούν και όλες αυτές οι συνεδριάσεις και συναντήσεις δεν έγιναν ποτέ. Αυτά είναι τα μαθήματα που πρέπει να συναχθούν από την ηφαιστιακή έκρηξη. Ευχαριστώ και επακούμε σε αυτό. Autant, UE, autant, c'est vrai. C'était une question de la présidence, quand même. <laughs> oui. Ναι, ναι, ήταν για τον ΝΑΤΟ, το θέμα της Προεδρίας, βέβαια, ασφαλώς. θέμα είναι ότι δεν θα επιληθούν βραχυπρόθεσμα ορισμένα από τα προβλήματα. Η κυρία Άστον, ο κύριος Ράσμουσεν, είπαν ότι θα συναντιούνται για να συζητούν και με τις ομάδες. και θα αναπτύξουν πιο αποτελεσματικά τις, τα θέματα των ικανοτήτων, την συνεργασία μας στο Αφγανιστάν με τον ΝΑΤΟ για να συμπληρώσουμε τα όσα πράττει το ΝΑΤΟ. διότι βεβαίως μπορεί να εκπαιδεύει απλούς αστυνομικούς ε, το ΝΑΤΟ όμως, όμως δεν εκπαιδεύει τους αξιωματικούς της αστυνομίας. Αυτό το για να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό χρειάζεται και μια εις βάθος συνεργασία και ανάλυση της κατάστασης. Το ίδιο και για την Αταλάντη. Δεν έχουμε δηλαδή ασφαλίσει πρόοδος προς το τι μπορούμε να κάνουμε μαζί. Για το πρόβλημα της συνεργασίας, του συντονισμού στη συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το Βερολίνο Plus, συν, που θεωρώ πως λειτουργεί. Αρκεί όμως, δεν είμαι σίγουρος. Έχει αποδείξει αποτελεσματικότητα μεν, αλλά και όρια το Βερολίνο Plus. Τα όρια τα είδαμε στη Βοσνία, δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες προτάσεις μεταξύ των οποίων ήταν να φτιάξουμε ένα επόμενο στάδιο του Βερολίνου Plus και μετά βεβαίως τον συντονισμό των δυνάμεων. Να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε την υπέρβαση, αν θέλετε, σε αυτό το σχέδιο συνεργασίας. Και τι είδους βούληση επιδεικνύουν τα διάφορα κράτη, κυρίως τα πιο δύσκολα, και πάντως από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί υπάρχει μια μικρή, μικρή, μικρή χώρα που έχει προβλήματα και μια πολύ μεγάλη χώρα του ΝΑΤΟ που έχει προβλήματα επίσης. Επίσης, σε ένα μέρος αυτής της μικρής, μικρής, μικρής χώρας έγιναν κάποιες εκλογές που άλλαξαν την ισορροπία στη διελκυστή των δυνάμεων. Και βλέπουμε νέα ονόματα, πρόσωπα που δεν γνωρίζαμε και θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσει η κατάσταση τώρα στο επόμενο διάστημα. Θα δούμε όμως στην πράξη. Και σας διαβεβαιώνω ότι υπάρχει βούληση μεταξύ του Γενικού Γραμματέως και της ΥΠΑ της Είναι στρατευμένη σε αυτήν την υπόθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρεσβευτά και το χρόνο σας σεβαστήκατε και στα θέματα δώσατε απαντήσεις πολύ ενδιαφέρουσες. Τα κύρια θέματα νομίζω τα κλείσαμε. Ένα μόνο για, το, για την ενημέρωση από τον Ρόμπερτ Κούπερ. Αύριο θα τον δούμε στην ΑΦΕΤ. Ε, θα έλεγα προλάβατε την ημερησία μας διάταξη. Όχι αύριο, δεν τον έχουμε δει ήδη. Πάντως ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Και από τον συνάδελφο κύριο Σφόποντα, ένα θέμα που έχει να κάνει με την Κίνα και την ασφάλεια. Επισημένω και εγώ ότι είναι πολύ μεγάλη σημασία στο θέμα και ελπίζω να το δούμε στην Επιτροπή μας σύντομα. Σε συνεργασία δε με τον ε, συνάδελφο Πασκού ε, ανέλαβα πρωτοβουλία για να ε, επικοινωνήσω με τις κινέζικες αρχές. Και έτσι όταν θα έχουμε την ευκαιρία στην υποεπιτροπή μα να μιλήσουμε για την Αταλάντη, για την Σομαλία κτλ. Θα προσκαλέσουμε και Κινέζους να μα μιλήσουν για τι προοπτικές και τι θέσει του. Πιστεύω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Προσβευτά. Κάνουμε ένα πολύ πολύ στομό διάλειμμα πριν περάσουμε στο επόμενο μας θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι η έκθεση για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής παρακολούθησης.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 Η συνάδελφος ε, Μαρία Ελένη Κοπά είναι υπεύθυνη, μας συζήτησε συγγνώμη, μα ενημέρωσε πω δυστυχώ σήμερα ε, λόγω ανωτέρα βίας δεν θα είναι παρούσα. Όμως, τη απουσία τη η Άννα Γκόμε θα μας παρουσιάσει την γνωμοδότηση. Ναι, Πρόεδρε, είναι η γνωμοδότηση της Μαρίας Ελένη Κοπά. Έχετε την γνωμοδότηση για την ε, έκθεση που μα έρχεται από την Ήτρε. Η Μαρία Ελένη θα ήθελε να υπογραμμίσει κάποιες ιδέες για την ενδιάμεση αναθεώρηση του προγράμματος ε, για την δορυφορική πλοήγηση όσον αφορά την αξιολόγηση της υλοποίησης, μελλοντικές προκλήσεις και τις προπτικές χρηματοδότησης. Υπογραμμίζω ότι το ένα είναι σημαντικό πρόγραμμα για την Ένωση εφόσον ενισχύει την ασφαλειά της και το μικρόφωνο της ομιλήτριας κάνει διακοπές, δεν την ακούμε και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη δύο βασικά θέματα. Καταρχήν, τι διεθνεί επιπτώσει ε, του προγράμματος και την πραγματικότητα που εξορισμού ε, λέει ότι καμία διαστημική πολιτική δεν μπορεί να διεξάγεται χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους υπόλοιπους φορείς ε, του τομέα. Γι' αυτό και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όσους ήδη δραστηριοποιούνται στην ε, δορυφορική πλοήγηση, να υπάρξει συνέργεια όσον αφορά τις τεχνολογικές πτυχές, αλλά και να διασφαλίσουμε τη συμβατότητα και όταν γι' αυτό είναι δυνατόν και την διαλειτουργικότητα ανάμεσα στα διάφορα συστήματα πλοήγησης. Όπω γνωρίζετε σήμερα το πρόβλημα της συμβατότητας σχετίζεται με το κινέζικο σύστημα Compass και με τις ε, κοινέ συχνότητε με το Γαλιλαίο. Η πρόσφατη ανταλλαγή επιστολών ανάμεσα στον πρόεδρο Παρόζο και τον Κινέζο Πρωθυπουργό έδωσαν ε, ε, κατέληξαν σε ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, αλλά όχι στη λύση του προβλήματος. Και γι' αυτό ζητάμε να σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις σχετικές ε, διαπραγματεύσεις. Το επόμενο πιο σημαντικό ζήτημα είναι να καταλάβουμε σε ποιο βαθμό το Γαλιλαίο αποτελεί καθαρά πολιτικού χαρακτήρα πρόγραμμα. Φυσικά η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν εξ αρχή πω το Γαλιλαίο είναι ένα πολιτικό σύστημα και υπό πολιτικό έλεγχο. Ωστόσο, επειδή αναγνωρίσαμε στην έκθεση Βόγκα του 2008 για την ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική, το Γαλιλαίο αποτελεί και πολύ σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις σε ΚΕΠΑ. Και η συνάδελφος Μαρία Ελένη θέλει να μα θυμίσει ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι ορισμένε υπηρεσίες του Γαλλίου, όπω για παράδειγμα οι δημόσια αριθμιζόμενε υπηρεσίες, είναι λεπτής διπλής χρήση, και αυτό σημαίνει την ανάπτυξη πιο συγκεκριμένων κριτηρίων ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνο ε, μη ε, εγκεκριμένων χρηστών. Γι' αυτό είναι σημαντικό να τονίσουμε πως όλοι οι χρήστε του Γαλιλαίου θα πρέπει να συμμορφούνται προς τον διεθνή νόμο, το χάρτη και τις διάφορες ειδικέ συμβάσει, ε, καθώς και τις συνθήκες της Ένωσης αλλά και τις κατευθύνσεις γραμμέ όσον αφορά τις εξωτερικές δράσεις της Ένωσης. Επιπλέον, εφόσον υπάρχουν τεχνικές δυνατότητε για να αποφευθεί η χρήση του Γαλιλαίου, για παράδειγμα από την διεύθυνση ε, πυράβλων, η κυρία Κοπά ζητά τη θέσπιση των απαραίτητων τεχνολογικών κριτηρίων όσον αφορά την δέσμευση των ε, δορυφόρων, λαμβάνοντα υπόψη ότι και τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη θα πρέπει να γνωρίσουν την ευαισθησία του προγράμματο όσον αφορά την εξαγωγή τεχνολογία, ιδιαίτερα για τα υλικά που συμπεριλαμβάνονται στην ε, ρύθμιση ένα Τέλος, υποστηρίζει ότι υπό καμία προϋπόθεση δεν θα πρέπει η ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική να συμβάλλει στη γενική στρατιωτικοποίηση του διαστήματος και τονίζει τις ευθύνες των φορέων στο διάσημο όσον αφορά την ε, ρήπανση και την ευθύνη τους σε περίπτωση ε, ατυχήματος. Η κυρία Κοπά τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη διεθνούς διαστημικού δικαίου και καλωσορίζει τον Ευρωπαϊκό Κώδικα για τις ε, δραστηριότητες ε, στο διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη της αν την ανάγκη περιορισμού των ε, καταλήπων και προτείνοντας τη δημιουργία ε, κάποιου νομικού μέσου. Τώρα, εκμεταλλεύομαι το γεγονός ότι έχω το λόγο για να σας πω εγώ ότι όταν εγκρέθηκε η έκθεση Φανφόγκαου για την Ευρωπαϊκή Διαστημική Πολιτική, πολύ εξημών στο Κοινοβούλιο θεωρήσαμε ότι και αυτή ήταν η άποψη γενικά σε αυτή την Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας, ίσως όχι σε άλλες επιτροπές οι οποίες είναι ιδιαίτερα αφοσιωμένες στο Γαλιλαίο και την πολιτική αποκλειστικά του χρήση αλλά εμείς είχαμε μια μεγάλη, έναν αντιπαράθεση όσον αφορά την χρηματοδότηση του Γαλιλαίου και εδώ σε αυτή την Επιτροπή ήμασταν της άποψης ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε πως παρά το γεγονό ότι δημιουργήθηκε ω πολιτικό σύστημα, είχε και στρατιωτικέ κρίσει και δεν μπορούμε αυτό το να αρνηθούμε και ότι ήταν και ανόητο να το αρνηθούμε. Ε, γιατί κάτι τέτοιο υποβάθμιζε τι δυνατότητε χρηματοδότηση που τελικά ξεπεράστηκαν και υποβάθμιση και τι δυνατότητές μας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Γι' αυτό νομίζω πως είναι σημαντικό να ξεπεραστούν με κάποιο τρόπο αυτές οι ε, απόψεις οι περιοριστικές. Και να δεχτούμε ότι υπάρχουν στρατιωτικέ σχέσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δεσμευόμαστε από τη συνθήκη και από το διεθνέ δίκαιο. Όχι, αντιθέτω. Αλλά επίσης πιστεύω πως αυτό οδηγεί σε ερωτήματα σε σχέση με τον αντίκτυπο, όπως λέει η Μαρία Ελένη, που έχουν άλλοι φορείς όσον αφορά την στρατιωτικοποίηση της χρήσης του διαστήματος. Δεν ξέρω αν έχουμε εδώ κανέναν που θα μπορούσε να μας απαντήσει. Αλλά θα ήταν σημαντικό κάποιος από το Συμβούλιο ή από οπουδήποτε να μας δώσει μια εκτίμηση θα έπρεπε να κάνουμε και μια αναθεώρηση της συνθήκης ε, για το διάστημα, ώστε πραγματικά να παρεμποδίσουμε την ε, χρήση την στρατιωτική. Στην, μάλλον την υπερβολική στρατιωτικοποίηση του διαστήματο. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Ε, βρίσκω τη γνωμοδότηση που προετοίμασε η Μαρία Έλενα. Θυμίζει όλε τι πτυχέ που ανέφερε. Είναι σημαντικό να τονίσουμε αυτή τη διάσταση υποστήριξης της ε, ΚΕΠΑ και αυτή την διπλή χρήση, διτή χρήση που μπορεί να γίνει, καθώς και όλες τις ε, ασφαλιστικές δικλείδες που θα χρησιμοποιήσουμε για να διασφαλίσουμε την ε, πολιτική χρήση και τον πολιτικό έλεγχο σε απόλυτη συμφωνία με τις συνθήκες. Κάποιος συνάδελφος θέλει να αντιδράσει σε σχέση με αυτή την γνωμοδότηση να προσθέσει κάποιο σχόλιο. Να δώσω το λόγο στην κυρία Καβαντά της Επιτροπής. Merci, Monsieur le Président. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω την ικανοποίηση της Επιτροπής για το πεδίο που καλύπτει αυτή η έκθεση, καλύπτοντας και προσδιορίζοντας κατά τρόπο επακριβή και εμπεριστατωμένο τα θέματα και τα ευαίσθητα σημεία του προγράμματος Γαλιλαίος. Ιδιαίτερα για τα 7 σημεία ιδιαίτερος του προγράμματος Γαλιλαίος. Θέλω να κάνω δύο παραπομπές. Καταρχάς, η πρώτη αφορά το σημείο 5, στο οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει στο εγγύς μέλλον πρόταση για, τις υπηρεσίες, για την υπηρεσία PRS, Και ελπίζουμε ότι οι προτάσεις αυτές, προτάσεις κειμένου, θα αποσταλούν στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από τι θερμέ διακοπέ, δηλαδή τέλη Ιουνίου, αρχά Ιούλιο. Για το δε σημείο 6, που είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη όλων των προγραμμάτων, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται πλήρω τι ανησυχίε που εκφράζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προς τις εξαγωγές ευαίσθητου υλικού, εξοπλισμού δηλαδή, σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό. Για τα πιο τεχνικά ζητήματα της κυρίας Γκόμες μου προσδιορίζει ο ειδικό μας σε ότι το υλικό GNSS και το ο Γαλλός προσδιορίζεται ότι θα υπάρχει η ότι θα ακολουθεί το Missile Technology Control. Είναι λίγο τεχνικά τα θέματα και ελπίζω να μπορέσουν να κάνουν δεκτή αυτή την απάντηση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές. Στην τεχνική ερώτηση κυρία Γκόμες, εγώ τίποτα άλλο δεν έχω να προσθέσω. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα την κυρία Κοπά. Είναι εξαιρετική έκθεση. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Διαρωτώ με βέβαια αν σε αυτό το πεδίο έχουμε ένα level playing field, ένα ισότιμο πεδίο δραστηριοποίηση. Ρεαλιστικά τώρα η, χρηματοδο... η χρηματοδότηση των εντολών για τον... την EADS τότε οι Ευρωπαίοι μόνοι που, έχουν, που υποβάλλουν προσφορές που μια ε, τέτοια συγχρηματοδότηση την προβλέπουν. Και θα λέγαω ότι είναι κάπως μη ρεαλιστικό να πιστεύει κανείς ότι εμείς μακροπρόθεσμα θα είμαστε καν σε θέση τις χρηματοδοτικές προϋποθέσεις να τις δημιουργήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε τεχνολογικά να είμαστε ανταγωνιστικοί και εμπορικά να είμαστε ανταγωνιστικοί χωρίς το θέμα της διπλής χρήσης dual use να μην το συμπεριλάβουμε. Όλοι οι ανταγωνιστές μας, κανένας από αυτούς δεν υπάρχει που να μην χρηματοδοτεί, ας το πω, δραστικά ε, προγράμματα ή εγχειρήματα άμυνας όσον αφορά τον στρατιωτικό αλλά και τον πολιτικό τομέα. Τίθεται εδώ το θέμα του Γαλιλαίου για μας και το θέμα της αντιπαράθεσης για παράδειγμα Κίνας και Ευρώπης ε, δεν διεξάγεται σε ένα ισότιμο πεδίο διότι οι Κινέζοι ιδιαίτερα μαζικά διασταυρούμενες χρηματοδοτήσεις ε, ε, διασφαλίζουν σε αυτό το εγχείρημα από πλευρά τους διτά. Και εδώ πρέπει να το δούμε κατά πόσο θα συμπεριλάβουμε αυτό το θέμα και το επιχείρημα, κατά πόσο θα είμαστε σε θέση μελλοντικά την δική μας πρωτοπορία τεχνολογικά να την διασφαλίσουμε και το τμήμα μας το 20% να το διατηρήσουμε στην παγκόσμια κλίμακα αν δεν υπάρξει αντίστοιχη χρηματοδότηση θα είναι χήμερα να διεξάγεται μια συζήτηση ε, και να απορρίπτουμε τέτοια χρηματοδότηση από την Ευρώπη και από την άλλη πλευρά να έχουμε ανταγωνισμό σε παγκόσμιο πλαίσιο που διασφαλίζει με αυτονόητο τρόπο την στρατιωτική συνιστόσα και έτσι αποκτά ένα τεράστιο πλεονέκτημα εμπορικά εναντί Ευχαριστώ. Θέλουν και άλλοι συνάδελφοι να λάβουν το λόγο νομίζω. Όχι. Καλώς. Τότε υπενθυμίζω τις ε, προθεσμίες για τις τροπολογίες προθεσμία 11 Μαΐου επανεξετάζουμε στις 2 και 3 Ιουνίου την βρομοδότηση της κυρίας Δοκοπά την υιοθετεί η ΑΦΕΤ στις 22-23 Ιουνίου η έκθεση που έχει αναλάβει η Ήτρε θα υιοθετηθεί στην Ήτρε στις 13 Ιουλίου και στην Ολομέλεια θα τη δούμε το Σεπτέμβριο. Εάν δεν υπάρχουν τις παρατηρήσεις, κυρίσω το πέρα στη συνεδριά σου και παρακαλώ τους συντονιστέ των ομάδων να μείνουν για το Προεδρείο. Παρακαλώ.